Bonjour, good morning, bon dia. Καλημέρα. Bonjour, good morning, bon dia σε όλους. Θα συνεχίσω μιλώντας πορτογαλικά. Ας ξεκινήσουμε τις σημερινές μας εργασίες βρισκόμαστε στο σημείο 4 ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτη πληροφορία. Έχουμε μεταξύ μας ε, σε αυτή την Επιτροπή ένα νέο μέλος. Ζουστίνα Βιτασκάιτ της ε, πολιτικής ομάδας Άλντε. δεν είναι παρούσα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να την καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Δεύτερη πληροφορία που θα ήθελα, δεύτερη ανακοίνωση. Συμπερίληψη στον κανονισμό του Κοινοβουλίου μιας πρότασης που αφορά το gender mainstreaming, την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου από τον βουλευτή αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΚΟ και τον, τον Αλφ Σβένσον και τον πρόεδρο της δικής μας Επιτροπής. Προτείνεται να συμπεριληφθεί μια πρόταση στον κανόνα 49. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα έγγραφο το οποίο μπορείτε να βρείτε μεταξύ των εγγραφών που σας έχουμε ε, διαθέσει. Αυτή η πρόταση θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτρόπων και στη συνέχεια στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Άλλη ανακοίνωση. αφορά το Συμβουλίο της Ευρώπης. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι Υπάρχει δυνατότητα από κοινού ε, συνεδριάσεων με το κοινοβουλευτικό δίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, χώρες, ε, ε, γυναίκες μάλλον χωρίς βία, έτσι ονομάζεται το δίκτυο αυτό. Δημιουργήθηκε το 2006 και διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Από το 2011 κύριος πρωταρχικός στόχος είναι η κύρωση της ε, συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση ακριβώς της βίας ε, κατά των γυναικών και της οικιακής βίας η επωνομαζόμενη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Μόνο η Τουρκία και η Αλβανία έχουν κυρώσει αυτή τη συνθήκη μέχρι στιγμής η διαδικασία κύρωση, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, στι κατοχώρε και στην Πορτογαλία. Ο εισηγητή είναι ο Μέντο Μπότα, ένα Πορτογάλο στο Συμβουλίο τη Ευρώπη. Και όπως είπα, έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε με αυτό το δίκτυο. Περνάμε στο σημείο 5, ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. συστάσεις των συνεδριάσεων της, της 6ης Νοεμβρίου και της 10ης Δεκεμβρίου. Τα έχετε λάβει ήδη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Σημείο 6. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 3ης Οκτωβρίου 2011. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και αυτά τα πρακτικά και περνάμε στο σημείο 7. Το σημείο 7 το οποίο αφορά την απαλλαγή 2011 για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Η συγγήτρια, η κυρία Κλειβέτη. Και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει να εξετάσουμε ταυτόχρονα και το σημείο 8, απαλλαγή 2011, Γενικός Προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκή Ένωση τμήμα 3, Επιτροπή. Δίνω το λόγο στην κυρία εισηγήτρια για τις δύο αυτές ε, εισηγήσει, η κυρία Κλειβέτη. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, συνεχίσω. θα ήθελα να μιλήσω ρουμάνικα, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε διερμηνία στη, ε, ρουμανική, από τη ρουμανική γλώσσα. Ίσως την επόμενη φορά να έχουμε. Για το σημείο 7, απαλλαγή 2011, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φίλων Όπως ε, φαίνεται, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η έκθεση, έχει πολλά νούμερα, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντική. Διότι κατά την άποψή μου αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ε, κάνει, επιτελεί ένα πολύ καλό έργο. Αφού διαβάσα το έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου, έκανα κάποιες προτάσεις στη γνωμοδότησή μου. Όσον αφορά το σημαντικό ρόλο του Ινστιτούτου αυτή για την πρόθεση της ισότητας των φύλων και της υποστήριξης της ενσωμάτωσης σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Τονίζω ότι οι στόχοι και οι καθήκον του Ινστιτούτου απαιτούν να διατηρηθεί ως ξεχωριστή εντότητα εντός του θεσμικού πλαισίου. Το 2011 ήταν το πρώτο πλήρες επιχειρησιακό έτος για το Ινστιτούτο από τότε που έγινε ανεξάρτητο οικονομικά και διοικητικά τον Ιούνιο του 2010. Οι ετήσιοι λογαριασμοί του, του Ινστιτούτου δείχνουν προϋπολογισμό σε ευρώ 7.530.000 για όλους τους τομείς η οικονομική του θέση από την 31η Δεκεμβρίου του 2011 και οι ταμιακές ροές και η λειτουργία για το ε, έτος 2011 του Ινστιτούτου συμφωνούν με τις διατάξεις του οικονομικού κανονισμού του. Επειδή το 50% ε, των συνολικών δεσμεύσεων μεταφέρθηκαν, θα ήθελα να ζητήσω από το Ινστιτούτο να κάνει προσπάθειες μείωσης των μεταφορών αυτών ε, σε αποδεκτά επίπεδα μεταφορών, ώστε να σέβεται την αρχή της ε, ετήσιας περίοδου. Επίσης, ε, θα ήθελα να εκδηλώσω την ικανοποίησή μου όσον αφορά τη δέσμευση του Ινστιτούτου για τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη βελτίωση των ε, accruals και όσον αφορά τη βελτίωση της, του ποσοστού απασχόλησης που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου. Θα ήθελα να καλωνορίσω την ε, έκθεση αξιολόγηση εκ των προτέρων που εστιάζεται στους στόχους και στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και τέλος θα ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητα τη δραστηριότητας προσέγγιση των φίλων του Ινστιτούτου και την ενεργό ε, συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις επειδή αυτό το ζήτημα ζητήθηκε να εξεταστεί επίσης και από τα πρόσφατα έγγραφα για την ισότητα των φύλων όπως η πρόταση οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ισορροπία των φύλων μεταξύ μη εκτελεστικών διευθυντών εταιριών που ε, υπάρχουν στο χρηματιστήριο, που είναι γραμμάρια στο χρηματιστήριο. Επίσης, ισορροπία φύλων στην ηγεσία των ε, επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αηφόρο ανάπτυξη. Ήθελα επίσης να προσθέσω ότι προσωπικά ε, βοηθήθηκα από αυτό το Ινστιτούτο, διότι όπω γνωρίζετε η Επιτροπή μα είχε μια αποστολή στο Δουβλίνο όπου εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να ζητήσω από το Ινστιτούτο κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση των δύο φίλων γενικότερα στο Δουβλίνο και τη ισότητα των φίλων στο Δουβλίνο και έλαβα γρήγορα όλες τις πληροφορίες που ήθελα και για όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής αυτής ε, πιστεύω αυτός θα ήταν ένας ενδιαφέρον τρόπο ενημέρωση. Ε, το να ρωτάμε δηλαδή το Ινστιτούτο να μας ενημερώνει για το έργο του όπως προτείνατε κυρία Πρόεδρε θα περάσω και στο σημείο 8 που είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ματρία Επιτροπή Απαλλαγή για το 2011 όπως γνωρίζουμε, δυνάμει του άρθρου 8 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόθεση της ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω το αίτημα υλοποίησης του προπολογισμού βάση φύλων σε όλου του ενδιαφερομένου δημοσιονομική διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που περιλαμβάνεται τώρα στην ετήσια έκθεση παρατηρήσει από το Ελεκτικό Συνεδρίο ή απαντήσει από την Κομισιόν που αφορούν δαπανέ σε σχέση με την προώθηση τη ισότητα γυναικών και ανδρών. Αντίθετα, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τι πολλέ παρατηρήσει του Ελεκτικού Συνεδρίου ή τι απαντήσει τη Επιτροπή όσον αφορά δαπάνε που σχετίζονται με την πρόθεση της ισότητας και από αυτή την άποψη ζητώ από το ελεγκτικό συνέδριο να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία εφόσον υπάρχουν σε σχέση με παρατηρήσεις που αφορούν δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Ταυτόχρονα θα ήθελα να κάνω έκκληση για περαιτέρω προσπάθειες ανάπτυξης δεδομένων ε, ειδικών για κάθε φύλλο που επιτρέπουν να παρακολουθούμε πώς οι δημοσιονομικές κατανομές επηρεάζουν τις επαγγελματικέ ευκαιρίες ανδρών και γυναικών και που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην έκθεση υλοποίηση του προπολογισμού. Το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί ευκαιρία να αναπτύξουμε και να εισάγουμε τέτοια δεδομένα και να υλοποιήσουμε τον προπολογισμό βάση φύλου ως εργαλείο για τη χρηστή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλειβέτη. Και τώρα ε, δίνω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, εάν κάποιο το, μέλος το επιθυμεί. Η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, μιλώ εκ μέρους της ε, σκιώδους του ΕΛΚ της κυρίας Ματερά, η οποία δεν μπόρεσε να ε, παρευρεθεί. Και θα ήθελα να συγχαρώ την, την κυρία Κλειδέτη για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Πρώτα απ' όλα για την απαλλαγή που αφορά στο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Η κυρία Ματερά συμφωνεί με την πρόταση της κυρίας Κλειβέτη, δηλαδή την χορήγηση απαλλαγής για το 2011. Και συμφωνεί επίσης και με την έμφαση και την υποστήριξη που παρέχει η κυρία ε, Κλειβέτη στην σημασία του έργου της, του Ινστιτούτου για την ε, πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων. Επίσης έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι το 2011 αυτό το οικονομικό έτος ήταν το πρώτο έτος κατά τη διάρκεια του οποίου το Ινστιτούτο λειτουργήσε διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητα είχε την ε, δυνατότητα να διεξάγει δικασίες πρόσληψης και σήμερα πλέον είναι πλήρως λειτουργικό. Ζητήθηκε επίσης να μειωθεί, να μειωθούν οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων του Ινστιτούτου έτσι ώστε να μην επαλληλευτεί το φαινόμενο που παρατηρήθηκε το 2011. Σημειώνουμε επίσης την σημασία του έργου του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Τώρα όσον αφορά το σημείο 8, το τμήμα 3 του Γενικού Προϋπολογισμού, η κυρία Ματερά θα ήθελε να σημειώσει ότι ως προς αυτό το σημείο είναι ε, ατυχές το γεγονό ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ισότητα των δύο φύλων. Παρά όλα αυτά, συμφωνεί με την κυρία Κλειβέτη ως προς αυτό που τονίζεται στο πρώτο, στην πρώτη παράγραφο της εισηγήσης της, της γνωμοδότησής της, ότι θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 8 να συμπληρωθεί και να αναφερθεί η πρόθεση της ισότητας. Τώρα, σε σχέση με το... την παρακολούθηση, θα πρέπει να βελτιωθεί αυτά που σας μετέφερα τώρα ήταν οι, απο, οι απόψεις της κυρίας και με την, Ματερά και με την άδειά σας κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω και τη δικιά μου άποψη πρώτον για το σημείο 7, για το Ινστιτούτο και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία κλιβέτη για την δουλειά που έκανε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα αυτό το ζήτημα είναι ακόμα πιο σημαντικό και Αμφισβητήθηκε η νομιμοποίηση του Ινστιτούτου. Ορισμένοι συνάδελφοι ζήτησαν την συγχώνευσή του με την, ε, υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι το Ινστιτούτο παρέχει μια προστιθέμενη αξία, ότι έχει μια σημαντικό ρόλο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να του ζητήσουμε να είναι πιο αποτελεσματικό και η ετήσια έκθεση που η οποία εκδίδει να, έχει, να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συνεργασία και πιο στενή συνεργασία με αυτό το Ινστιτούτο. Επίσης η διεξαγωγή ερευνών, στατιστικών ερευνών πιο συστηματικών, πιο επικαιρο... επικαιρών επικαιροποιημένων με στοιχεία πιο ε, νεότερα καθώς το, η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα υποβάλλει ε, την, έκθεσή της στην Επιτροπή, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να κάνει και το Ινστιτούτο. Θεωρώ ότι η ήδη στενή και επικοδομητική συνεργασία της Επιτροπής μας με το Ινστιτούτο θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα και η δουλειά του έργο, το έργο του Ινστιτούτου να γίνει πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό, αλλά επίσης και το έργο της Επιτροπής μας για την ισότητα των φύλων να γίνει πιο αποτελεσματικό. Άρα η θέση μου είναι βητή. Ναι, υποστηρίζουμε 100% το Ινστιτούτο, αλλά επίσης πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του και να οδηγήσει στην πρόταση, σε προτάσεις για συγκεκριμένα αχυροπιαστά ε, μέτρα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκαμπριά. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Λέτ. Κύριε Λέτ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, δεδομένου ότι το Ινστιτούτο ε, που εκπροσωπώ σήμερα μου δίνει τη δυνατότητα να δώσω το λόγο σε αυτό για να αναφερθεί πάνω στο θέμα. Για την απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις αιτίες μεταφοράς του 50% των συνολικών δεσμεύσεων. Ουσιαστικά το ετήσιο πρόγραμμα του Ινστιτούτου εγκρίθηκε το Φεβρουάριο, δηλαδή καθυστερημένα εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας. Αυτό έχει ως συνέπεια καθυστέρηση της δέσμευσης των κονδυλίων. Αυτή είναι η πρώτη αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι ότι κάποιες από τις μελέτες μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησαν δεν έλαβαν σωστές προφορές, ικανοποιητικές προσφορές όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει. Συνεπώς η δεσμεύση των χρημάτων καθυστέρησε. Και τέλος, όπως γνωρίζετε, το Ινστιτούτο παρέχει υποστήριξη στην Προεδρία του Συμβουλίου και όσον αφορά την Κυπριακή Προεδρία έλαβε πληροφορίες αρκετά καθυστερημένα το Ινστιτούτο όσον αφορά τον τομέα που έπρεπε να αναλυθεί. Αυτή, αυτές οι τρεις αιτίες ήταν εξωτερική κίνδυνη ουσιαστικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το Ινστιτούτο μέσα το 2011. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η μεταφορά στην λογιστική περίοδο των δεσμεύσεων. Αλλά για το μέλλον ε, θα προσπαθήσουμε να προβλέπουμε καλύτερα και θα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδου τα ζητήματα στο μέλλον. Όπω γνωρίζετε, βρισκόμαστε ακόμα σε πρωταρχική φάση και πιστεύουμε ότι θα ανακτήσουμε την ταχύτητα πορεία ε, φέτο. Ήθελα να σα περιγράψω τώρα την κατάσταση όσον αφορά και την τεκμηρίωση τη απογραφή ε, του φυσικού εξοπλισμού. Είχαμε δύο λάπτοπ τα οποία δεν είχαν αριθμό απογραφή και σύμφωνα με την πολιτική, η πολιτική μάλλον του Ινστιτούτου αυτή τη στιγμή έχει καθιερωθεί και έχει αναπτυχθεί σωστή διαχείριση των περιουσιακών μας στοιχείων και έχει εγκριθεί εσωτερικά. Έχουμε πλήρη τεκμηρίωση, επισήμανση και καταγραφή. Όσον αφορά τα ε, ε, χρεώσεις ακρού, ε, θα βελτιωθούν ε, βάσει των νέων λογαριασμών. Αυτές ήταν οι κύριες πτυχές που επισημάνθηκαν στην ε, διαδικασία, στην εκθεσία απαλλαγή όσον αφορά τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και του Κοινοβουλίου. Εμείς ως Ινστιτούτο αναμένουμε, προσδοκούμε να, εργαστούμε, να συνεργαστούμε στενότερα με σας την επόμενη χρονιά αναμένουμε ότι θα συντονίσουμε καλύτερα τις εργασίες μας με τις δικές σας και αν είναι δυνατόν να παριστάμεθα σε ορισμένες από τις συνεδριάσεις σας όπως το έχετε ζητήσει. Αυτό είναι το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών μας και επίσης αναπτύσσουμε και κάποιες μελέτες. Το 2013 θα είναι σημαντικό έτος για το Ινστιτούτο όπου αναπτύσσουμε το ευρετήριο ισότητα των φύλων και προβλέπεται να λάβει χώρα μια ε, τεράστια σύνοδος, πολύ σημαντική σύνοδος τον Ιούνιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές πτυχές ε, για τις οποίες θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στενότερα και το προσδοκούμε με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φερνάντες. Τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ναι. Στην εκπρόσωπο. Thank you very much, Juana uh, Justice. Ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπο τη Γενική Διευθύνση δικαιοσύνη σε σχέση με την, το οικονομικό έτος 2011 θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Επιτροπή δεν έχει σχόλια επί της ε, έκθεσης που υποβάλλεται στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, μια γενική παρατήρηση από τη γενική ε, παρατήρηση. Είμαστε ευτυχείς που το ελεγκτικό συνέδριο δεν διαπίστωσε καμία ατασταλία στην διαχείριση των οικονομικών Γενική Γενικής τη δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες. Η πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ah, sorry. Uh, Μάλιστα. Μιλούσε χωρίς μικρόφωνο. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κλειβέτη, ε, για να εκφραστεί. Μερικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ την συνάδελφο Γκαμπριέλ για την υποστήριξη για τις εκθέσεις που συντάσω, λέγοντας ότι είναι σημαντικές. Χαίρετε και ειλικρινά θεωρώ ότι εκπροσωπεί ε, αυτό κάτι θετικό για την ψηφοφορία. Επίσης να ευχαριστήσω τον, την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε που παληθεύουν, επιβεβαιώνουν το, το, θέμα για την απαλλαγή του Ινστιτούτου. Εγώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους ώστε που έχουν συμβάλει σε αυτό το διάλογο. Τώρα φυσικά αν υπάρχουν τροπολογίες θα για να θα μπορέσουμε να συντάξουμε μια πλήρη έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ την κυρία Κλειβέτη. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών στην Επιτροπή μας είναι 27 ε, Δεκεμβρίου, το μεσημέρι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο λοιπόν. Μέχρι με, πέμπτη μεσημέρι δηλαδή. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα 22 Ιανουαρίου. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού 18 ε, Ιανουαρίου θα συναντηθεί, θα υπάρξει ψηφοφορία και θα περάσουμε στην ψηφοφορία 18 Μαρτίου. Αυτές είναι οι προθεσμίες που πρέπει να έχει κάνει υπόψη του για αυτήν εδώ την έκθεση. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε και να περάσουμε στο σημείο 9 της για τάξεως μεταφορά στο Εθνικό Δέκιο και εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου 2004 κάθετος 113 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και παροχή αυτό. Η συγκίτρια είναι η κυρία Ζήτα Γκουρμάη, παρούσα, και θα της δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σε το συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά στην ε, Συνταγματική Επιτροπή έγινε συζήτηση για τα πολιτικά κόμματα και για το μέλλον τους και έτσι δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία να πω και εκεί την απόψή μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ε, να είμαστε πάλι εδώ. Πέρυσι το Δεκέμβριο όταν παρουσίασα το έγγραφο εργασίας ε, ελάχιστη όπως είχε προβλεφθεί. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η οποία ήταν απόλυτα διατεθειμένη να συνεργαστεί σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν την οδηγία 2014-113 καθώς ΕΚ, φυσικά αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην νομοθεσία ισότητα των φύλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ήταν πράγματι η πρώτη οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετώπισε το ζήτημα τη ισότητα των φύλων και τη διακρίση βάση φύλου εκτό του τομέα τη απασχόληση, Απαγορεύει την άμεση και την έμεση διάκριση βάση φύλου για στον τομέα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται ότι θα συνέτασε μια έκθεση υλοποίηση μέχρι τα τέλη του 2010 σύμφωνα με την οδηγία. Ωστόσο, μετά από πολλές αναβολές ενημερωθήκαμε ότι η έκθεση αυτή υλοποίηση ε, δεν επρόκειτο να συνταχθεί πριν το 2014 παρά το γεγονός ότι επανειλημμένω ε, διατύπωσα την ανάγκη και τόνισα την ανάγκη για ύπαρξη μιας τέτοιας έκθεσης ε, με πρόσφατα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά. Όπως γνωρίζετε, η αιτία που παρουσίασε η Επιτρόπη ήταν η συνέπειση του κειμένου ως έχει. Όπως γνωρίζετε, η ECG, η ε, ε, Ένωση Καταναλωτών, έθεσε τέλος ε, στην, περίοδο, στη, περίπτωση του τέστασα οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν μεταβατικές περιόδους ενός έτους που θα τελειώσει 21 Δεκεμβρίου 2012. Εκεί άλλαξαν ε, οι προτεραιότητες του δικαστηρίου όσον αφορά την ασφαλιστική εταιρεία και συζητώντας με την Κομισιόν επί του ζητήματος κατέστησε ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο δεν προλάβαιναν πια να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα. επίση εξήγησαν ότι οι αλλαγές για τον ασφαλιστικό τομέα ε, καθιστούσαν πρόεμοι την ύπαρξη έκθεσης ε, υλοποίηση ε, επειδή δεν υπάρχει αυτή η έκθεση ούτε ενημερωμένα δεδομένα σε σχέση με το, σημερινή κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη-μέλη στην έκθεσή μου τονίζω τι προτεραιότητε τι οποίε πρέπει να εστιαστεί η Κομισιόν για να εντοπίσει τα υπάρχοντα κενά και να προσδιορίσει λύση για την κάλυψή του. Έτσι λοιπόν ε, είχαμε μια συνάντηση και κάποια συμφωνία για αυτά και η Επιτροπή με ενημέρωσε ότι τώρα ξεκινούν ανταλλαγή πληροφοριών με τα διάφορα κράτη-μέλη. Αποτελεί λοιπόν μια καλή ευκαιρία να βεβαιωθούμε ότι θα προσέξουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. επίση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μα ευχαρίστησαν που το έγγραφο εργασία ήδη παρέχει κάποιε κατευθυντήριε οδηγίε. Τώρα, όσον αφορά τι συστάσει, σε περίπτωση αναθεώρηση τη οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα μέσα μαζική ενημέρωση και τη διαφήμιση. Δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν όσον αφορά την εκπαίδευση, τη δημιουργία, τη διατήρηση ε, διαφορών στερεοτύπων βάσει των φύλων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ακριβώ να αξιολογήσουμε τι συνέπειες του κειμένου έχει παρόλο που η αύξηση του κόστους είναι αναπόφευκτη. Αυτό σημαίνει ότι η συνεχής διάλογος μεταξύ της Κομισιόν και των ασφαλιστικών εταιριών πρέπει να συνεχιστεί ώστε να αξιολογηθούν οι συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Η απόφαση για το τεστ ΑΣΑ είχε αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα ότι ενώ η προσφυγή έγινε για αποφυγή της διάκρισης τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση για τις γυναίκες διότι ε, σημαίνει θα κοστίζει περισσότερο για τις γυναίκες ασφάλεια από ότι για τις άντρες. Αυτό πρέπει να το παρακολουθεί η Κομισιόν στενά. Επίση, πιστεύω ότι το θέμα της νομικής αβεβαιότητας δεν έχει αντιμετωπιστεί μέσω των δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών και χρειάζεται κάποια στιγμή αναθεώρηση της οδηγίας ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ε, πλήρες πληροφορίες και αξιόπιστα δεδομένα είναι επίσης ε, πολύ σημαντικά. Αναμένω περισσότερη διαφάνεια από την Κομισιόν όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση. Η καθιέρωση μιας σωστής βάσης δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας που σχετίζονται με τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την προστασία των θυμάτων διακρίσεων λόγω φύλου. Τέλος, η έγκαιρη μεταφορά τη οδηγία είναι επίση ουσιώδη σημασία και αυτή είναι η άποψή μου. Η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρω την εξουσία τη για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη για αυτή τη μεταφορά και όπω κατάλαβα είναι διατεθειμένοι να το πράξουν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Ζόλταν που παρενέβη και μα ε, βοήθησε εξαιρετικά. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την ε, εξαιρετική σα δουλειά και για τη γυναίκα σας που θα κάνει παιδί. Επίσης συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρουμάη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Η σκιώδη γητριά μα η κυρία Σκρίλευσκα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γι' αυτό θα μιλήσω εξ ονοματό τη. θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα σημεία. Ευχαριστή την κυρία Κουρμά για την, το έργο της, την προετοιμασία αυτής της γνωμοδότησης. το ζήτημα της ασφάλισης επισημαίνει, καθώς επίσης και το γεγονό ότι δημιουργείται μια δυσμενής κατάσταση η οποία μέσω των κατευθυντηρίων οδηγιών θα μπορούσε να γίνει καλύτερη για τις γυναίκες. Κατά την άποψή μου, εδώ χρειάζεται να έχουμε μια προσέγγιση κατά περίπτωση και φυσικά να μην βασιζόμαστε στα στερεότυπα για το ρόλο των ανδρών και των γυναικών. Τα οποία προφανώς οδηγούν σε δυσμενείς διακρίσεις κατά των γυναικών. Θεωρεί επίσης ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα ανασφάλεια δικαίου και από αυτή την έννοια χαιρετίζω την... το μήνυμα που αποστέλουμε στην Επιτροπή, την, την έτοιμά μας να αναθεωρήσει αυτή την οδηγία. Έθεξα και χθε το ζήτημα του ποιο είναι ο ρόλο των φορέων για την ισότητα το έθεξα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πλέον ευνοούμενη ε, Ευρωπαία. Ε, δεν, δεν βλέπω ακριβώ πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι φορείς για την ισότητα θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα για την εφαρμογή της νομοθεσίας, βοηθώντας τις γυναίκες που επιδιώκουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους και την ισότητα, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει. Φαίνεται πως αυτοί οι φορείς για την ισότητα καλύπτουν και ασχολούνται με άλλα θέματα. Και εδώ ζητούμε, συζητάμε αυτά τα ζητήματα στις Επιτροπές Λίμπες, στην Επιτροπή για την Εργασία. Και δεν γνωρίζω πώς ακριβώς μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά πιστεύω πως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο Αυτή της έλλειψη ανάληψη ευθύνη, αυτής τη έλλειψη εργαλείων, δεν έχουν στην διάθεσή τους ίσως τα κατάλληλα εργαλεία για να ε, βοηθήσουν τις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα και ώστε, ώστε τελικά να εφαρμοστούν νόμοι. Ε, αυτή είναι η άποψη της ε, κυρίας Σκριλευσκά και θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που θα της δοθεί να υποβάλει τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπάουερ και δίνω το λόγο στην κυρία Κριστίν Τομπόη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και για τις συστάσεις που μας είναι χρήσιμες στα πλαίσια του έργου που έχουμε και εμείς Λίγα λόγια μόνο για την, τελευταία χρονιά που, όπου αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα φυσικά. Σε, όπως ξέρετε, η οδηγία, η έκθεση μάλλον της Επιτροπής που προβλέπεται στην οδηγία 2004-113 επέβαλε στην Επιτροπή να δώσει έμφαση κυρίως στον τομέα της ασφάλειας λόγω των εξαιρέσεων που υπήρχαν ε, σε αυτό το τομέα. Και στην εφαρμογή προβλέπονται ειδικέ ε, διατάξεις. Ε, τίθεται τέρμα σε αυτές τις εξαιρέσεις στη πιθανότητα των, ε, των ασφαλιών να κάνουν ε, οι ατομικές ε, ατομικά ασφάλιστρα και φάνηκε ότι είναι απαραίτητο το 2011 να εγκρίνουμε κατευθυντέρειες γραμμές για τους ασφαλιστές αλλά και για τις χώρες μέλη και μέχρι το τέλος της, αυτής της χρονιάς να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Αλλά σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να εγκρίνουμε κατευθυντήριες γραμμές από πριν, πριν να φτάσουμε στην προθεσμία η οποία έχει επιβληθεί από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλη της εβδομάδας τελειώνει αυτή η προθεσμία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με αρχές ε, του 2013 τι θα κάνουμε? Θα δούμε όλες τις νομοθεσίες των χωρών μελών, να επαληθεύσουμε ε, το θέμα των εξαιρέσεων, πώς έχει, αν έχει τεθεί τέρμα, ποιες είναι οι διατάξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και το 2013. Αυτή η χρονιά θα μας επιτρέψει επίσης να δούμε όλη την εξέλιξη ε, σε αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό το λόγο το 2014 θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια έκθεση που θα μας δώσει μια σφαιρική εικόνα ε, ξεκάθαρη για το τι έχει γίνει και πώς έχουν τα πράγματα εν γέννη, διότι προσπαθ την, ε, αυτή τη δεμή κάνουμε μια επαλήθευση όλων των διατέξεων ε, της ε, 2004. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και. Τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο εκ νέου στην συγγετριά μας, την κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, ιδίως αυτά που αφορούν στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οδηγία αυτή επέφερε σημαντικές αλλαγές στην, στην αγορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να που η Επιτροπή δημιούργησε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μπορούν να συνεργάζονται με μια έτσι, ικανή ομάδα και να παρέχουν νομοθετικές προτάσεις. Είναι σημαντικό να το πράττουν και να δημιουργούν τέτοια έγγραφα όπως αυτή η γνωμοδότηση. Χρειάζεται να είμαστε μαχητικοί, πρέπει να το επιδιώξουμε αλλά επίσης μας δίνεται και δυνατότητα να, να επανεξετάσουμε τις θέσεις μας. Γι' αυτό ζήτησα και η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι τον Ιανουάριο, γιατί ήθελα να είμαι σίγουρη ότι όλοι ε, που θα προτείνουν τροπολογίες θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν διαβάσει την ε, γνωμοδότηση ή δυνατόν στην γλώσσα τους. Πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους σε, όσον αφορά αυτήν την ειδική περίπτωση, την περίπτωση την υπόθεση Τεστασά. Δυστυχώς, πολλά κράτη-μέλη στρέφονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Χρειάζεται ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει μια κοινή ανακοίνωση. Αποκινούμε την Επιτροπή ε, Ισότητας των Δύο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας ότι υπήρχε δυνατότητα εξαίρεσης, αλλά αυτή ήταν δυνατότητα. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιο κράτος μέλος να την επιλέξει την εξαίρεση ή θα μπορούσε και όχι. Και το θεωρώ αυτό υποχρέωσή μας δεδομένη στις κρίσεις δημοκρατικής νομιμοποίησης που ε, υφίσταται αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη. Δεν θα θέλαμε το μήνυμα προφανώς της Επιτροπής να είναι αγαπητέ γυναίκες θα πληρώνετε ψηλότερα ασφάλιστρα και πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητε ε, επικοινωνίας και δημοσιότητας και από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή για να στείλουμε προ τα έξω ένα μήνυμα ότι σεβόμαστε τις ίδιες τι αξίες μα. Και δεδομένου ότι ε, έχει τιμηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Νόμπελ Ειρήνη, αυτό συμπεριλαμβάνει όλους και όλοι, όλους όσοι βρίσκονται στο, στην αίθουσα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επιδείξουμε την προσήλωσή μας στις αρχές μας και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τη σκιώδη συγγήτρια. Χαίρομαι την... που άκουσαν την παρουσία της κυρίας Μπάουερ. Και ευελπιστώ ότι στο τέλος θα από... θα, θα σταλεί αυτό το θετικό μήνυμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σα ε, ευχηθώ καλά Χριστούγεννα γιατί θα πρέπει να φύγω από την αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Κουρμάη. Τώρα για να ολοκληρώσω τις προφορίες ε, που έχουμε ήδη δώσει για το χρονοδιάγραμμα προθεσμία υποβολής τροπολογιών 15 Ιανουαρίου στις 5 ε, το απόγευμα ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών 18 ή 19 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Απριλίου 2013. Μετά από αυτή την ενημέρωση λοιπόν Ας περιμένουμε να πάει 10 η ώρα για να αρχίσουμε να μιλάμε για το σημείο 10 ο κύριος Γκούσταυσον θα προεδρεύσει διότι και εγώ πρέπει να απουσιάσω για να πάω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επειδή από τις 10 προβλέπεται να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και ελπίζω να σας ξαναδώ όλους στις αρχές του νέου έτους με όλη την ενέργεια που θα χρειαστούμε για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας.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 ξαναρχίζουμε αρχίζουμε λοιπόν και φτάσαμε στο σημείο 10 το οποίο είναι μια παρουσίαση από τον εκπρόσωπο του UNFPA η κυρία Σίτσκε Στένεκερ Χαιρόμαστε που την έχουμε εδώ πέρα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Καταλαβαίνω ότι για την Επιτροπή μας αυτό το θέμα είναι προσφυλές. Δεν θα πω περισσότερα. Καλύτερα να σας δώσω αμέσως το λόγο και σας ευχαριστώ ξανά που είσαστε εδώ μαζί μας. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερο ευτυχή που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή και θα σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, η κατάσταση του παγκοσμίου πληθυσμού το 2012 που φέρει τον τίτλο «Κατόπιν επιλογής και όχι κατά τύχη». Αυτό γιατί επιχειρηματολογεί, εκθέτει το επιχείρημα ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τον αριθμό των παιδιών που θα κάνει κάθε πότε, ε, το, πότε θα, τα, θα κάνει παιδιά και να έχει πρόσβαση σε μέτρα αντισύλληψης. Το ανθρώπινο δικαίωμα λοιπόν στον οικογενειακό προγραμματισμό είναι ένα δικαίωμα το οποίο ίσως το θεωρούμε δεδομένο στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά όπως θα διαβάσετε και στην έκθεση δεν ισχύει κάτι τέτοιο για ολόκληρο τον κόσμο. Πανηλημένα ε, διασκέψεις έχουν αναφερθεί στην σημασία του οικογενειακού προγραμματισμού. 22 εκατομμύρια άνθρωποι, γυναίκες στο, στον, ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν πρόσβαση σε, στις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού αλλά ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες, σε ορισμένες ε, κοινωνικές ε, ομάδες όπως η οι ε, φτωχοί, οι έφηβοι, η τα μέλη των μειονοτήτων διαπιστώνουμε υψηλό αριθμό ανεπιθύμητων κήσεων. Η πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό μπορεί να περιορίζεται από έλλειψη χειραφέτησης, από τη φτώχεια, από διακρίσεις. Αυτές, αυτά τα προσκόμματα υποσκάπτουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Η πρόσβαση όλων των γυναικών στον οικογενειακό προγραμματισμό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, να συμπεριληφθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη στο κύριο σύστημα υγείας, να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τα δικαιώματα των, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και η καταπολέμηση των κοινωνικο παραγόντων που δίνουν το πρόβλημα. Η πρόσβαση στην οικογενειακό προγραμματισμό είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα οικονομικό και κοινωνικό μέτρο. Είναι οικονομικό το ζήτημα υπό την έννοια ότι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη δημιουργεί προβλήματα κοινωνικά, μπορεί να, μπορεί να καταστήσει το κορίτσι, ή τη γυναίκα ε, θύμα ε, μιας ε, διαρκώς επιδενούμενης κατάστασης, φτώχειας και αποκλεισμού. Οδηγούμαστε σε μια καταπάτηση άλλων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Γιατί μια γυναίκα η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή της. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζοντας το ζήτημα βοηθάμε τις γυναίκες να έχουν καλύτερο εισόδημα, καλύτερη εκπαίδευση και τελικά καλύτερη θέση και στην οικογένειά τους και στην κοινωνία. Έχει υποδειχθεί μέσω μελετών ότι ο οικονομικός προγραμματισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη. Η επένδυση στον οικονομικό προγραμμα... οικογενειακό προγραμματισμό αλλάζει την δομή του πληθυσμού ως προς τις ηλικίε ε, των μελών του πληθυσμού και μελέτες στο Μεξικό και σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι μειώνοντας τον αριθμό των εξατόμενων μελών σε μια οικογένεια μπορεί να έχει τεράστιες ε, σημαντικές και θετικές συνέπειες στην ε, κοινωνία και στην οικονομία. Οποιαδήποτε επένδυση χρημάτων προς αυτή την κατεύθυνση τελικά βοηθά τις οικογένειες, βοηθά την κοινωνία. Τα βασικά γεγονότα, τα βασικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν μαζί με το σχετικό φύλλο, τη σχετική έκθεση φέτος δείχνουν, αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ χαμηλής ε, αναπαραγωγής και της αναπαραγωγικής υγείας. Τα κυρία αποτελέσματα που βλέπουμε είναι ότι η επένδυση στον οικογενειακό προγραμματισμό και την αναπαραγωγική υγεία βελτιώνουν όχι μόνο την υγεία αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Η επενδύση στον οικογενειακό προγραμματισμό είναι μια μέθοδος στρατηγική αποτελεσματική ως προς το, κόστο. Ως προς το κόστος. Πολλές γυναίκες πεθαίνουν κατά την γέννηση, κατά την κοίηση με τον προγραμματισμό μειώνεται η θνησιμότητα των μητέρων κατά δύο τρίτα. Σήμερα ο οικογενειακός προγραμματισμός σε αναπτυσσόμενες χώρες κοστίζει δύο δισεκατομμύρια ετησίως και κατανέμεται μεταξύ κατοικιών, κυβερνήσεων και δωρητών. 8,1 δις το χρόνο θα κόστιζε αυτή τη στιγμή στις χώρες ο οικογενειακός προγραμματισμός, είναι το διπλάσιο αυτό, αλλά αυτή η πρόσθετη επένδυση των 4,1 δισεκατομμυρίων δολάριων θα εξοικονομήσει χρήματα τα οποία θα δαπανώνταν διαφορετικά σε υπηρεσίες για τις μητέρες και τα νεογέννητα το 2012. Το ε, διάφοροι οργανισμοί διεθνώς διοργάνωσαν μια σύνοδο κορυφής για δεσμεύσεις ώστε να γίνει διαθέσιμος ο οικογενειακός προγραμματισμός σε επιπλέον 130 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε αναπτυσσόμενες χώρες ως το 2020. Ο Άντερ Σπίλμπαξ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανάπτυξη, παρέστη στη Σύνοδο και υποστήριξε 23 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον υποστήριξη για, την για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Κάνοντας αυτή τη δέσμευση, ο Επίτροπος είπε ότι το να βοηθάμε τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις για το μέλλον. Στο σημερινό κόσμο όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το μέγεθος των οικογενειών τους. Αυτό αφορά την πρόθεση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και την προστασία της υγείας των γονέων και των παιδιών. Η Σύνοδο Κορυφή αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τον οικογενειακό προγραμματισμό και σημαντικέ πολιτικέ και οικονομικέ δεσμεύσει από δωρετέ όπως και από αναπτυσσόμενες χώρε. Όλε αυτέ οι εξέλιξει είναι πολλά υποσχόμενε, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα για να εξαλείψουμε τα προβλήματα και να επιτρέψουμε σε όλου να ασκούν το δικαίωμά του για οικογενειακό προγραμματισμό. Ευχαριστώ. Επόμενη διαφάνεια. Τι πρέπει να γίνει η κατάσταση το 2012 όσον αφορά τον παγκόσμιο πληθυσμό οι βουλευτές ε, οδηγούν τους ε, τα κοινοβούλια και διάφορους ενδιαφορεμένους να κάνουν τα εξή. Πρώτα απ' όλα να αυξήσουν την οικονομική υποστήριξη και την πολιτική δέσμευση ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει προγραμματισμός οικογενειακός διαθέσιμος σε όσους τον θέλουν, όποτε τον θέλουν και ότι οι υπηρεσίες, οι παροχές και οι πληροφορίες θα είναι υψηλής ποιότητας. Δεύτερον, η προώθηση του οικογενειακού προγραμματισμού ως δικαίωμα η άσκηση του οποίου επιτρέπει την επίτευξη ε, της εκπλήρωσης πολλών άλλων δικαιωμάτων. Η ενσωμάτωση του εθελοντικού οικογενειακού προγραμματισμού σε ευρύτερο κοινωνικό ε, προγραμματισμό και ανάπτυξη, διότι ο κοινωνικό προγραμματισμό βοηθάει και τα δύο, εξάλληψη των οικονομικών, κοινωνικών και οικονομικών ε, προσκομμάτων για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Όποιο λοιπόν το επιλέγει, επιλέγει τον προγραμματισμό αυτό, έχει πρόσβαση σε αυτό. Μείωση του αριθμού των ανεπιθύμητων ε, κοιήσεων και εκτρώσεων, βελτιώντα την αξιοπιστία και την ποιότητα τη αντισύλληψη και των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού οικογενειακό προγραμματισμό να έχει προγράμματα διαθέσιμα σε μεγάλο εύρος χρηστών όπως έφηβοι, άγαμοι και όσοι άλλοι το επιθυμούν. Και τέλος, δέσμευση ε, και συμμετοχή αντρών και νεαρών αγοριών στον οικογενειακό προγραμματισμό για την υποστήριξη των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών για τη χρήση αντισύλληψη. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ το πρόγραμμα δράσης που συμφωνήθηκε στη Διεθνή Σύνοδο του 1994 που έλαβε χώρα στο Κάιρο καθοδήγησαν ε, το έργο του Σχετικού Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών ώστε κάθε κοίηση να είναι επιθυμητή, κάθε γέννηση να είναι ασφαλής και να εκπληρώνονται οι δυνατότητες κάθε ατόμου. Στην 20η επέτειο του προγράμματος δράσης ε, το 2014 του προγράμματος δράσης του ΚΑΕΡΟ και τις προθεσμίες για τις NTG το 2015, οι κυβερνήσεις έχουν ανανεώσει τη δέσμευσή τους για το σχετικό πρόγραμμα δράσης και ζήτησαν από το UNFPA να διεξάγει συνολική αναθεώρηση των επιτευγμάτων, των κενών και των προκλήσεων για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος δράσης. Ταυτόχρονα αναθεώρηση της προόδου προς το NTG και θα συζητηθεί μια νέα συνένεση για την ανάπτυξη για την επόμενη γενιά. Για το μέλλον θα αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξη ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε ε, αναπαραγωγική υγεία και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα, οι συζητήσεις ε, για το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 όσον αφορά αυτή την ατζέντα μετά το 2015. Ελπίζουμε ότι εκεί θα υποστηριχθεί όλο αυτό. Η σύνοδη του 2013 της ε, Επιτροπής για την ε, κατάσταση των γυναικών που θα λάβει χώρα το Μάρτιο και ε, η Σύνοδος για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο θα ενταχθούν επίσης σε αυτόν τον διάλογο. Όσον αφορά τη διασφάλιση της οικουμενικής πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την υποστήριξη των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, απαιτείται ε, ε, πολιτική και οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότητα των φύλων, η ανάπτυξη των ανθρώπων θέτουν αυτό το ζήτημα στον πυρήνα των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση. Οι γυναίκε σε ολόκληρο τον κόσμο υπολογίζουν στην υποστήριξή μας. Δεν πρέπει να τι απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο για ερωτήσεις. Η κυρία Γκαμπριέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Στένεκερ για την παρουσίασή της. Απλώς να επανέλθω σε δύο-τρεις πτυχές να, να κάνω ενδεχομένω ερωτήσεις. Πρώτον, χαιρόμαστε που έχουμε αυτού του είδους τις εκθέσεις που μας επιτρέπουν από τη μια να αντιμετωπίσουμε τι είναι απαραίτητο να γίνει ε, και θεωρώ ότι το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τα διαφορετικά δεδομένα που έχουμε είναι η βάση που αποτελούν για να μπορέσουμε να έχουμε βέλτιστες πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ε, διαδίδονται, να ενημερωνόμαστε για αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, γιατί είναι θετικό. Επίσης, δίνω έμφαση σε μια από τις συνέπειες που είπατε υπάρχει σχέση ανάμεσα στον προγραμματισμό των οικογενειακό και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι πραγματικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα είναι πολύ ευαίσθητες όσον αφορά αυτό το επιχείρημα. Δεύτερον, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε είναι απαραίτητο να έχουμε πιο πολλά προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές είναι να δώσουμε έφαση στις μικρότερες ηλικίε. πριν να φτάσουμε δηλαδή σε ηλικίε όπου τα κορίτσια γίνονται μητέρες. Όσον αφορά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε έφαση στον εικονιακό πραγματισμό, έχω κάποιες εφυλάξεις για τον τρόπο τον οποίο μπορεί να γίνει έχοντας την εμπειρία από τις αναπτυσσέμενες χώρες και δει την Αφρική, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους επιβληθεί απ' έξω. Πρέπει να γίνει από μέσα. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση από τις ε, κατατόπων κυβερνήσεις. Όλες οι προσπάθειες από το ΝΟΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν περιορισμένα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν αυτό ε, κεντρικό σημείο να υπάρξει μια θέληση, μια προσπάθεια, αλλά θα πρέπει από μέσα να τους ευαισθητοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις χώρες να μπουν στο, στην ψυχή αυτή του προβληματισμού. Υπάρχουν ε, φυσικά διαφορετικές πολιτικές, δημόσιες πολιτικές φυσικά. Εδώ έχουμε επιχειρήματα, έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, ε, την ε, σεξουαλική ενημέρωση, ε, ξέρουμε ότι αυτά είναι θέματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ιδιωτικού χαρακτήρα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα θέματα. Τώρα, ερώτηση. Καλώς. Πρόσβαση όσον αφορά την πρόληψη, ενημέρωση, αλλά σίγουρα τίθεται το θέμα των οικονομικών μέσων. Εγώ πήγα στη Ζάμβια, όπου ο οργανισμός έκανε κάποιες μελέτες και έχει εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα ε, ε, να τους διώσουν, να τους ενημερώσουν, να τους δώσουν προφυλακτικά. Ε, θα έπρεπε να γίνει δωρεάν αυτό για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση και να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση. Αυτό το προβληματισμό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για αυτές τις χώρες. ξέρουμε ότι υπάρχει ε, η θέληση. Δεν είναι ότι δεν έχουν συνείδηση τη καταστάσεω, αλλά δεν έχουν τα μέσα. Δεύτερο ερώτημα. Οκ. Είναι θέμα στο οποίο πρέπει να ενταχθούν και οι άνδρες, τα αγόρια και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ε, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι χωρίς τους άνδρες, ειλικρινά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ε, θα ήθελα πιο συγκεκριμένα, ίσως κάποια συγκεκριμένα ε, παραδείγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. το λόγο στην κυρία Μωρή Σαρτιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που συμπεριλάβατε στην ημερήσια διάταξη εργασιών μας αυτό το θέμα. Όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορούμε να μοιραστούμε. Το μόνο που με λυπεί είναι ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μας δεν βρίσκονται εδώ για να το απολαύσουν. Διότι Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω. Έχουμε και μεγάλη πολιτική κινητοποίηση να κάνουμε για αυτό το ζήτημα. Υποστηρίζω τα όσα είπε μόλις η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ για τη συμμετοχή τελικά όλων των ενδιαφερομένων, όλων των μελών της κοινωνίας, των ανδρών, των νέων, ε, αγοριών σε αυτή την εκπαίδευση. Αλλά από πολιτική άποψη γνωρίζετε ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί πραγματικά ένα ζήτημα ενίοτε ταμπού. Ευχαριστώ λοιπόν που το εντάξατε στο πρόγραμμά μας, αλλά πραγματικά ένα ε, ζήτημα που προκαλεί διαφωνίες Στα όσα είπατε κύριε Διευθύντρια όσον αφορά την περιγραφή της πραγματικότητας και την αναλύσή σας είπατε ότι το να αναγνωρίζετε το δικαίωμα στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία σημαίνει κύρωση και άλλων δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι σήμερα δεν πρέπει να διαχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Για εμάς, από πολιτική άποψη, πρέπει να κινητοποιηθούμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες, έτσι ώστε η αναγνώριση του δικαιώματος ε, στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία να αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της ε, αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω και επίσης ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι σημειώνεται σταθερή πρόοδος επί του θέματος. Εγώ είμαι Γαλλίδα. Είναι ένα θέμα αυτό που η Σιμών Βέιλος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε προωθήσει στη Γαλλία το 1975. Δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 35 χρόνια που τέθηκαν σε αυτά τα ζητήματα στη Γαλλία. Και η Σιμών Βέιλ ήταν μια γυναίκα μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρατηρούμε ακόμα και σήμερα ότι διαρκώς πρέπει να προσέχουμε ώστε να έχουμε κατά συνείδηση ψηφοφορίες επί του θέματος ώστε αυτό το ζήτημα να μπορέσει να προχωρήσει. Προωθώντας αυτό το ζήτημα προωθούμε ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν λοιπόν εντάξετε αυτό το θέμα της αναπαραγωγικής υγείας στα ανθρώπινα δικαιώματα θα μας βοηθήσετε πολιτικά να προχωρήσουμε. Και αν δεν προχωρήσουμε θα οπισθοχωρήσουμε. Αν οπισθοχωρήσουμε εδώ, οπισθοχωρούμε παντού. Προσοχή λοιπόν. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό τα κεκτημένα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι ότι υπάρχει μια σχέση που υπογραμμίσατε εσείς μεταξύ της γεννητικότητας και της ε, αμοιβή των γυναικών. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυριότερα μας αφορά η ισότητα των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, των αμοιβών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνοχή σε αυτόν τον προγραμματισμό ώστε να προωθήσουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την ισότητα της αμοιβή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ ο ίδιος θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, για τις οποίες απαντήσετε. Σκέφτηκα σε αυτά που είπατε μας δείξατε και εικόνα ότι πόσο ε, ε, αποτελεσματικό μπορεί να είναι στο θέμα με το κόστος για τις οικογένειες. Ε, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι επενδύει κανείς σε κάτι και κερδίζει κάπου αλλού. Καμιά φορά προσαρμόζεται κανείς. Γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Όταν επενδύει κανείς ένα δολάριο, αφού είναι γνωστό ότι θα αποδώσει κάτι παραπάνω, γιατί είναι τόσο γρήγορο να ληφθεί μια απόφαση. Ουσιαστικά δεν θα έπρεπε αυτό καν να το βλέπουμε σαν κόστος. Είναι μια επένδυση. Δηλαδή τα χρήματα θα επιστραφούν. Γιατί όμως είναι τόσο δύσκολο για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις να το κάνουν. Το άλλο ερώτημα. Εσύ τι πιστεύεις κάτι για συγκεκριμένο στην Ευρώπη, ε, στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Πώς, πώς ξέρει, εσύ ξέρεις για κάποια, ποιες είναι οι δυνατότητες, αλλά έχεις υπάψη τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και να είναι αποτελεσματικό εδώ στο Κοινοβούλιο. Και τρίτον, σε σχέση με αυτά που είπε η συνάδελφος, το να επιβάλλει κανείς στις άλλες χώρες ε, απ' έξω Ανέφερε εσύ ότι πρέπει να έρχεται από μέσα. Το σέβομαι αυτό που λες, συνάδελφε. Για μένα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν μιλάει κανείς για αυτά. Δε, πολλές φορές το κάνει κάπω να έρχεται από πάνω να επιβάλλει κάτι. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Καταλαβαίνω την προβληματική. Είναι όμω συγκεκριμένο το ερώτημα σε σχέση με αυτό. Πάρα πολλέ χώρε. Ε, έχουν υπογράψει την σύμβαση για τις γυναίκες και έχουν καθήκον να κάνουν κάποια θέματα σε αυτόν εδώ τον τομέα. Σε αυτά τα πλαίσια δεν θα έλεγαμε κανείς ότι ε, ε επιβάλλει κάτι. Θα ήθελα ειλικρινά να δω σε σχέση με το ερώτημα σε, ε, σε, τη συναδέλφου, δηλαδή το να, πώς ανταποκρίνονται οι χώρες σε αυτά που προτείνουμε. Λοιπόν, όλε αυτέ οι ερωτήσει είναι αρκετέ. Μπορείτε να δώσετε και την απάντησή σα. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ σημαντικά σημεία που θέτετε και τις πολύ ενδιαφέρουσε ε, ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επανέλθω στα όσα είπε η κυρία Γκαμπρίελ. Συμφωνώ απόλυτα. Το επιχείρημα, το οικονομικό είναι εξαιρετικά πιστικό. Και παρότι πολλοί από εμάς ε, θα θεωρούσαμε ότι ο οικογενειακό προγραμματισμό είναι ένα δικαίωμα πρωταρχικά, το οικονομικό επιχείρημα είναι εξαιρετικά έγκυρο και πιστικό και όπως τόνισε και ο πρόεδρο. Για κάθε δολάριο που επενδύουμε στον οικογενειακό προγραμματισμό εξοικονομούμε 1,40. και Όπως λέτε λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι τόσο δύσκολο ορισμένες κυβερνήσεις να αντιληφθούν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έλεγε ουσιαστικά ότι έχουμε έλλειμμα οράματος εδώ. Ότι είναι κοντόφθαλμο το όραμα των πολιτικών. Και φυσικά έχουμε και περιορισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες και εκεί υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά, ανταγωνιστικές συνιστώσεις που πρέπει να ερευνηθούν αλλά θα θέλαμε πραγματικά να κάνουμε έκκληση για να υπάρξει αυτή η μακροπρόθεσμη, το μακροπρόθεσμο όραμα και να αντιληφθούμε ότι πέραν όλων των άλλων ωφελών που επιφέρει ο οικογενειακός προγραμματισμός στις γυναίκες, στους άντρες, στις οικογένειες και στις χώρες υπάρχει και ένα απτό οικονομικό όφελος. Αναφέρατε επίσης ε, ένα πολύ σημαντικό σημείο ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση σεξουαλική ανάλογα με την ηλικία και αυτό φυσικά θα προσαρμόζεται στο πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρα, κάθε κοινότητα. Αλλά πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αυτό που είπατε για τη συμμετοχή των αντρών είναι πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα μια χώρα όπω ο Νίγερα. Μια πολύ ευάλωτη χώρα έχει την υψηλότερη γονιμότητα στον κόσμο. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες αποκτούν 7 παιδιά σχεδόν. Η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια ήταν περίπου 2% ετησίως και η ανάπτυξη του πληθυσμού 4% ετησίως. Αν κάνει λοιπόν κανεί τι μαθηματικέ πράξει και τα υπολογίσει, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ευάλωτη χώρα με ελάχιστη αρδεύσιμη γη έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ποιότητα της ζωής θα υποβαθμιστεί αντί να βελτιωθεί. Το 1 τρίτο μόνο των παιδιών πηγαίνουν στο σχολείο, το 1 τέταρτο των κοριτσιών μόνο πηγαίνει στο σχολείο. Η κατάσταση απαιτεί δράση. Και αν δούμε και το τι αρδεύσιμη γη υπάρχει σε μια χώρα όπως τον Νίγηρα, τώρα έχουν περίπου πληθυσμό 15 εκατομμύρια, το 2015 θα έχουν φτάσει στα 50 εκατομμύρια το 2050 και δεν θα υπάρχει καθόλου αρδεύσιμη γη. Πρέπει να γίνει κάτι λοιπόν και η ίδια κυβέρνηση του Νίγηρα πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάτι και τα τελευταία δύο χρόνια άρχισαν πραγματικά να το αντιλαμβάνονται και να αναλαμβάνουν δράση. Μία από τις δράσεις που κάνουν ε, για να συμμετέχουν οι άντρες, γιατί φυσικά μιλάμε για ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον, πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Τι έκαναν λοιπόν. Έχουν σχολεία για συζύγους άντρες, όπου οι σύζυγοι, οι άντρες, μαθαίνουν διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων την αντισύλληψη και το δικαίωμα των συζύγων, γυναικών τους, στο να έχουν άποψη ως προς το πόσα παιδιά θέλουν να αποκτήσουν. Δεν είναι εύκολο, ειδικότερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα που αναφέρατε ότι η σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία ορισμένες φορές ε, ε, αντιμετωπίζεται ως ταμπού. Αληθεύει. Εμένα δεν μου είναι πάντα κατανόητο. Πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλές παρανοήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτό θεωρώ είναι ένα από το καθήκον του UNFPA να απομυθοποιήσει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ότι ουσιαστικά αυτό αφορά το δικαίωμα των ανθρώπων να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν πότε, πώς και κατά πόσο θέλουν να αναπαραχθούν. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 ουσιαστικά άρχισε να αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα. Και ε, επαρελειμμένα αναφέρεται και μερικές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί στις διαπραγματεύσεις αποτελεί τόσο δύσκολο ζήτημα όπως είπατε, πράγματι αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα που θα βοηθήσει την υποστήριξη όλων των άλλων δικαιωμάτων που θέλουμε να απολαμβάνουν οι γυναίκες. Δεν είναι λοιπόν σωστό, πιστεύω, να είναι τόσο αντιφατικό αυτό το ζήτημα ορισμένες φορές. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε όσον αφορά τον αντιφατικό του χαρακτήρα. Η Επιτροπή για την Κατάσταση των Γυναικών θα λάβει χώρα το Μάρτιο, αφορά τη βία κατά των γυναικών. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες η Γενική Συνέλευση, η τρίτη Επιτροπή της Γενικής συνέλευση υιοθέτησε ένα πολύ προοδευτικό ψήφισμα για τη βία κατά των γυναικών και εκεί αναφέρεται επίσης και η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και το δικαίωμα των γυναικών που έχουν υποστεί βία και σεξουαλική βία ότι και αυτές έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες ε, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ειδικευμένε. και ε, πιστεύω ιστορικό, ιστορική ένδειξη είναι ότι αναφέρονται και τα αναπορικά δικαιώματα σε αυτό το ψήφισμα. Ε, αναμένουμε λοιπόν αυτή την Επιτροπή για την κατάσταση των γυναικών και δεν βλέπω να υπάρχει λόγος για τον οποίο το CSW δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει κάτι παρόμοιο. Αυτέ είναι δύο σκέψει που είχα να κάνω για αυτό το ζήτημα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάρα πολλά πράγματα. Κατά πρώτον, όπως επισήμωνα και το αναφέρει και πολύ καθαρά η έκθεση, τα χρήματα εξακολουθούν να αποτελούν ένα ζήτημα. Δεν έχει λυθεί το να κατανείμουμε λοιπόν επαρκα... επαρκή κονδύλια στο ζήτημα της σεξουαλικής και αναπορικής υγείας και ειδικότερα στον οικογενειακό προγραμματισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να καθοδηγήσει την πορεία για την περίοδο μετά το 2015, τα ETG, SDG, όπως και να ονομάζονται. Όλοι αυτοί οι στόχοι που καθοδηγούν αυτές τις συζητήσεις για το πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015 πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβεβαιώσουμε ότι η οικουμενική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική αγία θα βρει τη θέση της σχετίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό με την ισότητα των φίλων και τα δικαιώματα των γυναικών που πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να μεριμνήσουμε να εκπροσωπείτε επαρκώς σε όλους αυτούς τους διαλόγους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε που ήσουν εδώ πέρα. αυτό που, με το οποίο δουλεύουμε εμείς εδώ πέρα είναι ε, δηλαδή η δική μου προοπτική είναι ε, το να προστατεύσουμε το σώμα της γενεϊκάς σημαίνει να την προστατεύσουμε να βγει στην κοινωνία, στην αγορά. Έχουν, το βασικό θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές φορές μπορεί να φυσικά να δημιουργούν αντιπαραθέσεις. Συμφωνώ ότι είναι. Μπορεί να είναι δύσκολο να έχει κανείς τον πλευρό του σε αυτά τα θέματα και τους άνδρες. Θα το κοιτάξουμε. Καμιά φορά δίνεται μια έμφαση ότι η, τα δικαιώματα των γυναικών είναι κάτι άλλο από ανθρώπινα. Αν το βλέπανε έτσι ότι τα δικαιώματά τους είναι ανθρώπινα δικαιώματα και οι άνδρες θα ήταν διαφορετικά. Αλλά δεν γίνεται. Ε, δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση ε, απλώς από την ανδρική πλευρά είναι σαν να βάζει στην άκρη το μισό πληθυσμό και λέει φροντίστε μόνοι σα τα δικά σας θέματα. Ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε αυτές τις απόψει. Χρειάζονται κατάρτιση και οι άνδρες. πολύ μάλιστα. Τέλο πάντων. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι οι περισσότεροι που είναι σε θέση να πάρουν μια απόφαση, αποφασίζουν, έχουν εξουσία, είναι άνδρες. Δεν είναι τόσο πολλές οι γυναίκες. Οι άνδρες λοιπόν ενδιαφέρονται περισσότερο αυτοί οι άνδρες από τα χρήματα. Η δική μου προσέγγιση όσον αφορά το οικογενειακό πραγματισμό έχει κοινωνική πτυχή και οπτική γωνία, αλλά είναι σημαντικό συχνά να μιλάμε και για τα λεφτά, την οικονομική πτυχή. Πρέπει να σκεφτούμε. Αν σκέφτεται κανείς ότι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται στο δικό μου γήπεδο να παίξουν, ε, θα πάω στο δικό του, Θα το δω από τη σκοπιά του χρήματα, επένδυση κτλ πραγματικά να του δείξει κανεί, κοιτάξτε αυτό είναι επένδυση. Ίσως έτσι όλοι αυτοί οι άνδρες που βρίσκονται σε θέση ισχύω και εξουσία να μπορέσουν να ε, έρθουν στα νερά μα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Και θεωρώ δηλαδή, προϋποθέτω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Καλώ uh, Καλώς. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση και πηγαίνουμε στο αυτό το έκτακτο σημείο που έχουμε σήμερα σε διάταξη. Draft oral question, etc. etc. Λοιπόν, για τη βία κατά των γυναικών και τα λοιπά. Αναγκάστηκα να, το, να πω δύο-τρία στα αγγλικά για να καταλάβετε που αναφέρουμε. Λοιπόν, ξέρετε το πλαίσιο η Επιτροπή μας προσπάθησε να κάνει μια, ένα ψήφισμα για το 16 ημέρες τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη για θέματα βίας κατά των γυναικών. Δεν τα καταφέραμε στην Ολομέλεια. Ε, αποφάσισαν οι συντονιστές στο Στρασβούργο να αποσύρουμε το ψήφισμα και να κάνουμε όπως είχαμε πει παλιότερα. Δηλαδή, να πάρουμε αυτό το ψήφισμα όταν η αντιπροσωπεία μας θα πάει στη Νέα Υόρκη στο... και τότε να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα ψήφισμα. Φυσικά να θέσουμε κάποια ερωτήματα στην Επιτροπή. Για να γίνει αυτό εφικτό και για να προλάβουμε χρονικά ούτω ώστε να έχουμε την, ε, το, το ψήφισμα, την απόφαση στο, στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Τι κάναμε. Οι συντονιστές μου δώσαν εντολή να κάνω μια πρόταση, πρόταση ψηφίσματος και ερωτήσεις και στη συνέχεια εσείς αφού του κάνετε κάποιες αλλαγές, προτάσεις, τροποποιήσεις τέλο πάντων, τροπολογίες, να προχωρήσουμε. Να σας πω ίσως γενικά τι ακριβώς, περί πρόκειται αυτή η πρόταση. Δεν είναι και τίποτα παράξενο. Στην πρόταση ψηφίμισματος που έχουμε, ας πούμε, λέει ότι συχνά μιλάμε στην Επιτροπή για Βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών και είναι ένα σφαιρικό παγκόσμιο πρόβλημα υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για, το, για, για τους οποίους γίνεται, αλλά το βλέπουμε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν δηλαδή προσδιορίζεται ιδιαίτερα σε ένα χώρο, σε μια τάξη. Ε, στα πλαίσια του We Are Us ε, ε, βλέπει κανείς το θέμα του, της βίας κατά των γυναικών και και πριν από 1,5 χρόνο στο Στρασβούργο το Κοινοβούλιο πήρε μια, έκανε ένα ψήφισμα και εκεί έχουμε υλικό. Επίσης στην πρόταση αναφέρεται ότι απαιτείται πολιτική θέληση για να γίνει κάποιο ουσιαστικό, κάποιο ουσιαστική πρόοδος. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν και φυσικά με μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, με κοινωνικές ε, δράσεις όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει να το δούμε, να είμαστε πιο ενεργοί ε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, να ενισχυθεί ο ρόλος και η δραστηριότητα όσον αφορά να, να δοθεί δηλαδή έμφαση και να προβληθεί αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Υπάρχει φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τα κονδύλια για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Δεν, δεν αξίζει να λέει κανείς ότι αυτά τα θέματα είναι σημαντικά, χρειάζονται πόροι, κονδύλια. Ωραία, ρητορικά μπορεί κανείς να λέει το α και το β. Δεν θα γίνει τίποτα αν δεν έχουμε και τα χρήματα που χρειάζονται για να δράσουμε. Κάτι άλλο είναι σημαντικό σε όλες τις περιπτώσεις να ενισχύσουμε το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και να δοθούν και κονδύλια και εκεί. Οι, οι UN Women το Ηνωμένων Εθνών οι γυναίκες είναι πολύ ενεργές και δραστήριες σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το έργο μας να δούμε μια προοπτική για την ισότητα. Αυτό να διακρίνει όλες τις εργασίες και σε συνεργασία με την υπηρεσία του, των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν συστάσεις των, ε, συστάσεις των υπερογνωμόνων για το λεγόμενο Global Implementation Plan, ένα πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την εφαρμογή αυτού, αυτά σε γενικές γραμμές στο κείμενο που έχουμε. Θα κάνουμε φυσικά κάποια ερώτηματα στην ε, Επιτροπή. Δεν προλαβαίνουμε όμως να το υποβάλουμε στο Συμβούλιο. Με αυτό σημαίνει ότι κάνουμε μια πρόταση, η τα μέλη μπορούν να, κάνουν, να κατασένουν τροπολογίες για αυτό το κείμενο και να αποφασίσουμε τον Ιανουάριο το, στη συνεδρίαση τότε μετά από αυτή την εισαγωγή δίνω το λόγο σε όποιον το επιθυμεί. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να πει, θέσει, να πει κάτι. Uh, Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την άποψη της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η συνάδελφός μου, γιατί η Επιτροπή συνεργάζεται συχνά, στενά με την ε, υπηρεσία αυτή για την προετοιμασία της θέσης μας. Της θέσης μας της CSW είναι μεγάλη τιμή για μας να απευθυνθούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει το έργο έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επιτροπή για, το, για την Κατάσταση των Γυναικών, την CSW. Επομένω, η συζήτηση μα σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη γιατί θα μα δώσει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίση είμαστε ευτυχεί που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκπροσωπηθεί με αντιπροσωπεία στη CSW. Όπω γνωρίζετε, η βία κατά των γυναικών είναι ένα δομικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα δεδομένο και η καταπολέμησή του αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώ. Φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα στρατηγικό πλαίσιο και ένα ε, πρόγραμμα δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένε δράσει με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. και την πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων. Ο ειδικό εισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει, όπως γνωρίζετε, προσφάτως αναλάβει καθήκοντα και είναι στις προτεραιότητές του η βία κατά των γυναικών. Ε, θα τον συναντήσουμε την, ε, του χρόνου στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του πάνελ υψηλού επίπεδου της SW. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την προσέγγιση της Επιτροπής για τις προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη χρονιά. Είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το γεγονός ότι η 57η φετινή CSW δεν κατάφερε να καταλήξει συμπεράσματα και αυτό μας έδωσε δύο διδάγματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρί, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κοινή θέση. τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίση πρέπει να ξεκινήσουμε νωρί να απευθυνόμαστε προ τα έξω στην κοινωνία των πολιτών. Όπω αναφέρατε κι εσεί, έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσει με τα κράτη-μέλη για την υιοθέτηση τη κοινή θέση, ήδη από το Σεπτέμβριο, και ευελπιστούμε ότι αυτέ οι συζητήσει θα ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα. Όπω γνωρίζετε, η επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρυφεί από την συλλογική μα ε, δράση και προσέγγιση από τις προσπάθειες όλων μας. Γι' αυτό προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, να αναλύσουμε τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα και οι στόχοι μας είναι δύο. Πρώτον, η, η ε, Επιτροπή για το Στάτους των Γυναικών την επόμενη χρονιά να καταλήξει συμπεράσματα και δεύτερον, να υιοθετήσουμε μια κοινή ε, προσέγγιση η οποία θα μας βοηθήσει να μην υπάρξει οπισθοχώρηση σε σχέση με, το, με τα ήδη κεκτημένα. Συνεργαζόμαστε με ομάδες, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Γυναίκες, ε, οργανώσαμε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες και συζητήσαμε με οργανώσεις γυναικών πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε την παρουσία μας στη CSW. Έχουμε προσπαθήσει επίσης να απευθυνθούμε τόσο σε χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιες θέσεις με τις δικές μας, αλλά επίσης και σε χώρες ε, με τις οποίες οι θέσεις μας διαφέρουν, γιατί αυτού του είδους η πυθό είναι απαραίτητη αν θέλουμε να καταλήξουμε στα συμπεράσματα του χρόνου. Χώρες της Λατινικής Αμερικής τον Ιανουάριο θα διοργανώσουν μια σύνοδο με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει το ζήτημα του φίλου. Ήδη σα ανέφερα τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να επιδιώξουμε συνεργασίες και να παραστούμε στη CSW. Επίση θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε παράλληλε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στη συναδελφό μου έτσι ώστε να δώσει, δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την, ε, το έγγραφο της θέσης της, Επιτροπής, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πέτρο. Βαδίνουμε τώρα το λόγο στην κύριε Φέστρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω δυο λόγια για το περιεχόμενο του εγγραφού θέσης το οποίο συντάσσουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν βασικές γενικές κατευθυντήριες αρχές και πιο συγκεκριμένες αρχές. Πρώτα απ' όλα σκόπος είναι φυσικά να έχουμε μια σταθερή δέσμευση υπεράσπισης ε, του κεκτημένου όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι το πρώτο. Και φυσικά δεύτερον να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις δεσμεύσεις. Δεύτερον, φυσικά να συνεχίσουμε να υιοθετούμε προσεγγίσεις βασισμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε συγκεκριμένες αρχές. Όπως το να λέμε ότι η βία κατά των γυναικών ε, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι είναι αδύνατο να αιτιολογείται καθιονδήποτε τρόπο η βία κατά των γυναικών. Δεύτερον, το να συσχετιστεί η βία των γυναικών με τη διακριτική μεταχείριση. Επίσης, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης. Επειδή, όπως γνωρίζετε, αυτό θα είναι ένα από τα κυρία θέματα φέτος, η προστασία των θυμάτων. Ο ρολός των ανδρών Επίσης θα υπερασπιστεί και θα προβληθεί έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ιδέα υποστήριξης και των στόχων της ε, χιλιετίας. Των και η σημασία παρακολούθησης του φαινομένου και ανάπτυξης ε, στατιστικών στοιχείων. σκόπος είναι να δούμε ήδη τι είναι σημαντικό σε αυτό το κείμενο και τις δεσμεύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Συμπεριλαμβανομένου και των μη κυβερνητικών οργανισμών και των δραστηριοτήτων τους. Σκοπός είναι να έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα με πολύ ισχυρέ δεσμεύσει. Και θεωρητικά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να χρειάζεται να μιλάμε για συγκεκριμένες μορφές βίας κατά των γυναικών, αλλά να προσπαθούμε να έχουμε μια γενικότερη προσέγγιση, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε μακροσκελή κείμενα που είναι πιο δύσκολο να διαπραγματευτούμε. Αυτό που προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε σε όλες τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη τα ε, ισχυρότερα κείμενα και τις ισχυρότερες δεσμεύσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, το να συμπεριλάβουμε αναφορές σε διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις που περιλαμβάνουν έγγραφα περιφερειακής εφαρμογής και διεθνείς δεσμεύσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη συνεργασία και τη στήριξη και άλλων κρατών σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Θα μπορούσα να διακόψω εδώ. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε. Θα μιλήσω σιωδικά, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι σε αυτά που είπατε. Η πρόταση που έχουμε, η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί, υπενθυμίζω. Είναι στα σημεία 8 και 9 για το λεγόμενο Global Implementation, Global Advocacy, Prevention of Violence, etc. Πάνω σε αυτό το θέμα. Έχετε συζητήσει ε, στα πλαίσια των εργασιών που κάνετε, έχετε κάποια θέση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε την απάντησή σας, αφού σας πήρε τόσο χρόνο να τη συζητήσετε. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν αναφερόμαστε στην εκστρατεία παγκοσμίας υπεράσπισης των δικαιωμάτων και δράσης. Αναφερόμαστε στην πρόβλεψη, στην πιθανότητα το 2015 να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δάση στο το Πεκίνο συν Και θα θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να ε, τελικά να καταλήξουμε σε αυτό. Έχουν ήδη ξεκινήσει ε, συζητήσει για το πώ τελικά θα καταλήξουμε στο Πεκίνο συνήκωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει και εκείνη τη συζήτηση πώ θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να διοργανωθεί, Πιθανώ όχι να διοργανώσουμε μια ε, διεθνή διάσκεψη η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πλατφόρμα δράση του Πεκίνου καθώ επίση και τα κεκτημένα ω προ την ισότητα των δύο φύλων ίσως ήταν πιο σκόπιμο να διοργανωθεί μια μεγάλη εκστρατεία μια εκστρατεία εορτασμού, ευαισθητοποίησης και απολογισμού των επιτευγμάτων που ήδη σημειώθηκαν. αναρωτιόμασταν εάν θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτήν την ιδέα που ε, έχει ε, κυκλοφορήσει καθώς επίσης με, την ε, παγκόσμια εκστρατεία στην οποία αναφέρεστε εδώ, την Global Advocacy Campaign. γιατί η μία ιδέα ίσως αποτελεί εξειδίκευση της άλλης. αυτή τη στιγμή προβάλλεται αυτή την ιδέα, θα θέλαμε να έχουμε κάποιε περισσότερε πληροφορίε, κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε σε σχέση με το τι, στο, στο τι συνίσταται αυτή η εκστρατεία. Όχι, δεν έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε για το Global Advocacy Campaign, αλλά γνωρίζουμε ότι α, είχε αφαιρθεί την πιθανότητα διοργάνωσή τη, ίσως να μπορούμε να τη συνδέσουμε με άλλη εκστρατεία, κατά τρόπο που εσείς θεωρείτε πιο πρόσφορο δεν έχω να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα είναι ανοιχτό το ζήτημα, το οποίο επίσης συνδέεται με το σημείο 8 περί του παγκοσμίου προγράμματος δράσης και η πρόταση για του συμπρογνώμονες είναι και αυτή μέρος, μέρος της, ε, του έργου σας. Ναι, η Επιτροπή επιβεβαιώνει. Συμμετέχει συμμετείχαν εκπρόσωποι μας στις διεργασίες που διοργάνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο, στο πλαίσιο της CSW και επίσης υπήρχε εκπροσώπηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο γιατί θεωρούμε σημαντική για την επιτυχία της διάσκεψης της CSW του χρόνου την παρουσία και την, την ε, συμβολή της ε, UN Women. Επανέρχομαι στα Σουηδικά. Ευχαριστώ λοιπόν για όλα. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα για αυτό το θέμα. Να υπογραμμίσω απλώς θα αποφασίσουμε ε, αφού του στείλω την πρόταση τροπολογίες προθεσμία είναι 12η ώρα 9 Ιανουαρίου η Επιτροπή 21 Ιανουαρίου θα ψηφίζει και πιθανότατα περνάμε στο Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Και με αυτά κλείνουμε με αυτό το σημείο. Επίσης να πω στην αρχή της ενεδρίασης είπαμε καλωσορίζουμε δύο ομάδες επισκεπτών. Να, τα να ξανακαλωρίσω αυτές, ε, αυτές, αυτές τις ομάδες που ήρθανε και τις δύο ομάδες ε, επισκεπτών τις καλωσορίζω εγκάρδια. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Περνάμε στο σημείο 11 τώρα. Αντίκτυπος οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των, ε, της γυναίκας. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, σημαντικό για την Επιτροπή μας. Έχουμε αποφασίσει ότι είναι το θέμα το οποίο θα είναι ε, το, ένα σημαντικό θέμα για την 8η Μαρτίου. Προσφυλές λοιπόν θέμα. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Μωρίν Σαρτιέ, να μας το παρουσιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που που ε, θέσατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής μας. Είναι μια έκθεση ε, στην οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε το σύνολο των πολιτικών ομάδων. Είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο μπορούμε πραγματικά να περάσουμε, να ενημερώσουμε στα πλαίσια της ημέρας της γυναίκας την 8η Μαρτίου και είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να κινητοποιήσουμε και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ξέρω, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης είναι αυτό το θέμα ε, υπομελέτη. Για, θα γλωμοδοτήσουμε συγκεκριμένα. Είμαστε εδώ σε ένα θέμα λίαν σημαντικό, διότι τελικά, από τη μια, την είναι ε, ένα υπόγειο θέμα σιωπηλό, και γιατί. Διότι η κρίση έχει μεγάλες επιπτώσεις στις ε, γυναίκες και δεν μιλάμε πολύ, για την απασχόληση εννοώ, και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ε, τόσο γνωστό. Δεν έχουμε πολλούς δείκτες. Γι' αυτό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ε, από, να ωφελθούμε από την δημοσιότητα που θα δοθεί την 8η Μαρτίου να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και το Ινστιτούτο του Βίλνιους που μελετά την ισότητα των φύλων ούτω ώστε να έχουμε στη θέση μας πρόσφατες στατιστικές και αξιόπιστες. Είναι λοιπόν ε, θέμα το οποίο είναι στην καρδιά του προβληματισμού μας γιατί την έχουμε την μια ισότητα ε, των ε, ατόμων αλλά και την απασχόληση, αλλά είναι ένα παραμελημένο θέμα, διότι οι επιπτώσεις στις γυναίκες όσον αφορά την κρίση είναι κάτι το οποίο περνάει σε δεύτερο πλάνο. Όλες οι μελέτες δείχνουν στον κόσμο ότι η απασχόληση των ανδρών σε, σε περιόδους κρίσεως είναι κάτι το οποίο θεωρείται προτεραιότητα. Γι' αυτό σε εμά έγκυται να δώσουμε, να ρίξουμε τα φώτα πάνω σε αυτό το θέμα. Και φυσικά στη μελέτη μας, εδώ στην έκθεση, υπογραμμίζουμε ότι η κρίση οδήγησε τις γυναίκες σε μια πιο ε, επισφαλή θέση όσον αφορά την απασχόληση. Διότι αυτές είναι ήδη που ήταν σε επισφαλείς ε, συνθήκες απασχόλησης. Το καθεστώς των γυναικών ε, οι φέρει πίν. τι ήταν, μερική απασχόληση, επισφαλής απασχόληση, περιορισμένε συνθήκε. Αυτά είναι για τις γυναίκες. Και είναι οι πρώτες θέσεις οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση. Το δεύτερο θέμα πάνω στο οποίο δίνουμε έμφαση είναι ότι οι γυναίκες δεν ε, δεν έχουν μόνο αυτές τις επιπτώσεις της κρίσεως. Ε, οι πρώτες θέσεις εργασίας που επλήγησαν από την κρίση είναι τη... ήταν ε, θέσεις στις οποίες κατά πρωτόρυτα αποσχολούνται άνδρες. Βιομηχανία, βαριά βιομηχανία. Οι γυναίκες πού είναι περισσότερο. Είναι περισσότερες σε διοικητικές θέσεις Ε, και από θέσει που βρίσκονται πιο πολύ στον δημόσιο, θα λέγαμε, τομέα. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές των χωρών μελών, όπου και εγώ φυσικά συμφωνώ παρόλο που ε, βλέπω τις επιπτώσεις που υπάρχουν στους προπολογισμούς των χωρών μέλων, διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές λιτότητος οδηγούν σε μια κατάσταση όπου ε, πλήττεται περισσότερο η γυναική απασχόληση. Εκεί είναι περισσότερες οι γυναίκες σε αυτόν τον τομέα, στο δημόσιο. Ένα τρίτο στοιχείο, σε περίοδο κρίσεως, αναφέρομαι σε στερεότυπα, έτσι, διάφορα κλισέ, τι διαπιστώνει κανείς. Δυστυχώς, παρόλα όσα μπορούμε να πούμε ισότητα πολιτών, ό,τι και να έχουμε κάνει για την ισότητα των πολιτών, τα στερεότυπα ισχύουν. Οι άνθρες και η απασχόλησή τους είναι προτεραιότητα και οι γυναίκες έχουν την τάση οι ίδιες, οι ίδιες να υποχωρούν από την αγορά εργασίας, σιωπηρά. Αποχωρούν σε περιόδους κρίσεως για να πάνε πού? Σε άτυπη εργασία, άτυπη απασχόληση, ή αμυσθεί να απασχοληθούν κάποιοι. Βλέπουμε λοιπόν ένα τρίτο σημείο το οποίο μας φαίνεται εξήλσου ε, δύσκολο και το οποίο θα πρέπει να πολεμήσουμε για αυτήν εδώ την περίοδο της κρίσεως. Τέταρτο. Να δώσω μια έμφαση στις ε, επιπτώσεις κρίσεως στους ε, μισθούς. Οι γυναίκες υποχωρούν προς ε, επισφαλής απασχόληση, ε, όχι καλά αμοιβόμενη, μερική απασχόληση και πραγματικά μπαίνουν σε, μια, σε ένα κατήφορο και θα οδηγήσει φυσικά στο να έχουν και λιγότερη μειωμένη σύνταξη. Βραχυπρόθεσμα υπάρχει ένα άμεσο, μια άμεση επίπτωση όσον αφορά την ε, ε, απασχόληση των γυναικών, αλλά η κρίση βλέπουμε ότι έχει μέσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ε, φτωχοποίηση θα λέγαμε των γυναικών. Μακροπρόθεσμα όταν θα φτάσουν στη σύνταξη. Και υπάρχουν τα στερεότυπα ότι η, επιμένω σε αυτό ότι η ανεργία των ανδρών είναι κάτι που είναι πιο σοβαρό και αυτό είναι βαθιά ριζωμένο. Κάτι που θα πρέπει να δούμε φυσικά στις πολιτικές που θα ασκήσουμε. Σήμερα ξέρουμε ότι η μείωση, το, η μισολογή για διάφορους λόγους, αυτούς που σας ανέφερα, οδηγούν σε μια μεγαλύτερη φτωχοποίηση των γυναικών, ε, κοινωνικό αποκλεισμό. Πάντα οι γυναίκες πλήττονται. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, για παράδειγμα, ε, οδηγούν σε μεγαλύτερη ε, δυσκολία για τη θέση των γυναικών για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν στην απασχόληση. Σήμερα στις μονογονικές ε, οικογένειες ε, βλέπουμε ότι η, η πλειοψηφία αυτών ε, ε γύρω από την, θα λέγαμε, τον γυναικείο πυλώνα και εκεί έχουν δυσκολίες να βρουν μια απασχόληση, να ε, βρουν κατοικία αλλά έχουν και το βάρος ότι έχουν τα εξαρτώμενα θα λέγαμε άτομα, τα παιδιά, ηλικιωμένους να φροντίσουν η κοινωνία μας λοιπόν είναι τέτοιοι οργανωμένοι που είναι η γυναίκα αυτή η οποία τους αναλαμβάνει. Αυτούς τα παιδιά, τους γονείς, ε, άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτά με τη συνέχεια, στη συνέχεια ευαισθητοποιούν τη θέση της γυναίκας. Επίσης, να επιμείνω σε ένα άλλο, ότι η κρίση οδηγεί σε μια αύξηση της άτυπης απασχόλησης σήμερα μετά από μελέτες του ΟΣΑ η άτυπη αντιπροσωπεύει 33% του ΑΕΠ των χωρών μελών του ΟΣΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε περίοδους κρίσης αναγνωρίζεται η αντιπεργασία. Έτσι, εκεί οδηγούνται οι γυναίκες. Εξωθούνται θα έλεγα. Κάτι ακόμα σημαντικό. Οι γυναίκες είναι τέσσερις φορές περισσότερες στην ε, μερική απασχόληση από ότι οι άνδρες. Και η άτυπη λοιπόν και η, ε, μερική απασχόληση είναι για τις γυναίκες. Άλλη, μεγάλη, άλλη τόση επιβάνηση για τη θέση των γυναικών. Κι όμως, κι όμως, όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι σε περίοδο κρίσεως μία ισότιμη ένταξη στην αγορά των ανδρών και των γυναικών θα ήταν ένας παράγος, παράγοντας συγγνώμη, μια μιας δυναμικής, μιας ανάπτυξης και δυνατής μάλιστα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Να να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και να δούμε ότι στην ημέρα των γυναικών εμείς να κάνουμε θέμα στο ότι σε περίοδο κρίσεως η γυναίκα ε, μπορεί να έχει ένα ε, δυναμικό ρόλο και αυτό είναι που θέλω εγώ να θίξω. Επίσης να υπογραμμίσω κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ, λίγαν σημαντικό οι ανισότητες οι μισολογικές ανάμεσα στους άνδρες και τις γενικές, τα έχουμε δει αυτά. Είδαμε τους λόγους ε, που οδηγούν ε, φυσικά σε άνηση μεταχείριση και ε, συμβάσεις, μερικές αποσχόλες. Αλλά σε περίοδο κρίσης οι γυναίκες δέχονται ακόμα μεγαλύτερη, πλήγονται ακόμα περισσότερο της τάξης στο 17% στις ευρωπαϊκές χώρες με αποκλήσει σημαντικές ανάμεσα στις χώρες, στις διάφορες. Όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αυτές οι αποκλήσει οι παρόλο που έχουμε να κάνουμε ενδεχομένω με ίσες, ίσα προσόντα, σε, ίσε θέσει, έχουν να κάνουν ότι οφείλονται στο ότι η γυναίκα έχει και το, την αναπαραγωγή, ότι θα γεννήσει παιδιά. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και μια τελευταία που έγινε από ο ΩΣΑ δείχνει ότι ένα παιδί σημαίνει 12% λιγότερο μισό για τη γυναίκα, για τη μαμά. Κάθε παιδί οδηγεί σε ένα μισό μείωση τάξη 12%. γυναίκα η οποία προσλαμβάνεται, έχει ίδια προσόντα με ένα άνδρα, παίρνει μια θέση ανάλογη με ενός άνδρα, ήδη έχει ένα μειωμένο αμισό 17% λόγω του ότι θα μπορεί να πάρει άδεια γονική ε, και βλέπουμε για κάθε παιδί υπάρχει αυτή η επόπτηση του 12% Πού θα καταλήξει αυτή η γυναίκα όταν φτάσει στη σύνταξη. Άρα, με την έκθεση θέλουμε να πούμε ότι προτείνουμε να δημιουργηθούν πολιτικές οι οποίες θα μειώσουν τις ανισότητες, αύξηση της απασχόλησης ε, των γυναικών ε, σε σχέση με τους άνδρες. Επίσης, ε, πόροι από του τους υπέρ των γυναικών να επαναδροσοποιηθεί η γυναίκα, να αναβαθμιστεί ο ρόλος της γυναίκας και να κοιτάξουμε να βοηθηθούν να προβληθούν τέτοιες πολιτικές Ξέροντας φυσικά ότι θα έχουμε κάποιο εμπόδιο, διότι η επιστροφή στο χώρο εργασίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκά Ταμεία δεν θα πετύχουν αν δεν λάβουμε υπόψη χρειάζεται η συνεχής κατάρτιση αν δεν κάνουμε όλες τις προσπάθειες προσπάθειε, όλε οι ενέργειε που χρειάζονται για να ξαναφέρουμε τη γυναίκα στην αγορά εργασία. Διότι έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν την επαγγελματική. Και προσέτουμε σε αυτά και την κατάρτιση. Ξέρουμε ότι αυτό θα αποτελεί ένα επιπλέον ε, εμπόδιο, ένα επιπλέον βάρος για τη γυναίκα. Και εδώ φυσικά πάλι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα στερεότυπα. Ε, ε, θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε μια έμφαση σε αυτό εδώ το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ε, η Γκουρμάγερ είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο και όποιος άλλος το επιθυμεί. Παρακαλώ. Mm, thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. πρώτα απ' όλα να πω είναι πάντα μεγάλη, χαρά να, μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με την Ελίζαμπε και τα σχόλια, η γνωμοδότηση που έχετε προετοιμάσει είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από την δικιά μας την πλευρά πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει η δημοσιοποίηση του ζητήματος. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εντός και εκτός κοινοβουλίου, Και θεωρώ σημαντικό λοιπόν που θα προετοιμαστεί μια έκθεση επί του ζητήματος. Όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, νομίζω το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό που ονομαζούμε ε, σιωπηρή κρίση. Οι πολιτικές λιτότητες τις αναφέρατε, οδηγούν σε καταστάσεις επισφαλούς εργασίας, αλλά η κρίση δεν είναι η μόνη που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά λειτουργήσε σαν επιβαρυντικός παράγοντας, ένας παράγοντας ο οποίος επιβάρυνε τις ήδη υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Μας ε, βοηθά ίσως να επισημάνουμε και να αντιληφθούμε την, το, την μισθολογική ανισότητα, τη δυσκολία των, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες να συμβιβάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, την ε, εργασία σε επισφαλή ε, μορφή ή με μερική απασχόληση κτλ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι υπήρξε μια αλλαγή κατά τη διάρκεια χρονικά της κρίσης. Αρχικά υπήρξε ένας πρώτος κύκλος τις οποίες ε, τις επιπτώσεις τις ένιωσαν πιο έντονα οι άνδρες, αλλά αργότερα όταν η κρίση επεκτάθηκε στον τριτογενή τομέα, όπως για παράδειγμα τον τραπεζικό, δεν λάβαμε υπόψη μα το γεγονό ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι ανάγκε εκείνου που πλήττεται εξαιτία τη απόλυση που, για παράδειγμα, θα, θα, θα ε, υποστεί. Για παράδειγμα, στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα των υπηρεσιών απασχολούνται πολλέ γυναίκε οι οποίε έχασαν τη δουλειά του εξαιτία τη κρίση. Χρειάζεται, χρειαζόμαστε πιο επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τον αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας στα δύο φύλλα οι πολιτικές λιτότητες ε, έχουν αρνητικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα ή σε μεγαλύτερο βάθο αρνητικό στις γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί μία πλήρης και συνεκτική στρατηγική. Καλωσορίζουμε επίσης την ε, υιοθέτηση της οπτικής του φύλου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική απασχόληση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης τις τοπικές αρδιωτερότητες κάθε κράτους μέλους, την ανάγκη για διαβίου μάθηση και επαγγελματική κρατάρτιση, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τομείου... καθώς επίσης και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες για την πράσινη οικονομία. Ορισμένες παρατηρήσεις επιπλέον. Αναφερόμαστε στην κρίση και στη λιτότητα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές επιπτώσεις. Η Ελίζαμπετ ανέφερε ότι η φτώχεια έχει γυναικείο πρόσωπο. Όντως οι γυναίκες ε, υφίστανται δυσμηνή αντίκτυπο της ε, κρίσης και της οικονομικής και αυτό που ανέφερα και πριν, της δημοκρατικής κρίσης. Επομένως πρέπει να θυμόμαστε ότι θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε ήδη στοιχεία που έλεγαν πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μισθολογικές ανισότητες των γυναικών, πώς θα φτάσουμε από το 50% στο 60% της απασχόλησης των γυναικών. Στη νέα στρατηγική για την Ευρώπη 2020 δεν έχουμε πλέον αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε έναν αριθμό, έχουμε ένα στοιχείο που λέει ότι πρέπει η απασχόληση να φτάσει στο 70% συνολικά στην αγορά εργασίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και άνδρες και γυναίκες. Αλλά στην πράξη τι συμβαίνει. Περισσότερο από 70% των αδρών απασχολούνται στην αγορά εργασίας, ενώ λιγότερο από 70% των γυναικών απασχολούνται. Και εδώ υπάρχει μια συνωμοσία σιωπή. Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι όταν υπάρχει ανεργία ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης τη είναι οι γυναίκες να μείνουν σπίτι. Διαφωνώ οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής. Αν θέλουν να επιλέξουν να παραμείνουν στο σπίτι τους και να φροντίσουν την οικογένειά τους, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Αν θέλουν να ε, μπουν στην αγορά εργασίας, έχουν επίσης το δικαίωμα να το κάνουν. Μιλάμε επίσης για την συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσία, στα διοικητικά συμβούλια κτλ. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια για οικονομική ανάκαψη. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η εκθέση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα στις ε, γυναίκες της καταπληκτικής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θυμόμαστε όλοι ότι όλοι μας θα πρέπει, θα λάβαμε μαζί το βραβείο Νόμπελ. Και είναι σημαντικό που συμμετέχουμε σε αυτή το πολύτιμο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, και σε όσους συμμετείχαν στην εκθέσή μου να ευχηθώ σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα στις 8 Μαρτίου εφόσον το αντιμετωπίσουμε πολύ επαγγελματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκαμπριέλ. Είπαμε, έχουμε ψηφοφορία 11 και 30. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι θέλουν να μιλήσουν. 11 και 30 θα κάνουμε διάλειμμα γιατί αυτό το έχουμε δηλώσει για την ψηφοφορία και μετά μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό ε, μην ανησυχείτε. Κύριε Γαβριέλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να χαιρετήσω την εισηγήτρια κυρία για την πολύ πλήρη παρουσίαση της εκθεσής της. Εγώ θα πω τα πράγματα κάπως καθαρά. Θέλουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια έκθεση ολοκληρωτική που θα μας επιτρέψει ως για πρώτη φορά να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που θα ενσωματώνει στο ίδιο κείμενο τα διάφορα συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε εντοπίσει και επισημάνει όλοι μας σε διάφορε εκθέσει. Αυτό ήθελα να προβάλλω, λοιπόν, το πιο σημαντικό σημείο, όπως θεωρώ εγώ αυτή τη έκθεση, που βασίζεται με πολύ επαγγελματικέ και ε, εύλογες ε, εύλογα επιχειρήματα ε, συμπεριλαμβάνει όλες τις πολιτικές που χρειαζόμαστε αυτή η έκθεση. Τρία σημεία υποστηρίζω την κυρία Συγήτρια όταν λέει ότι πρέπει να συζητήσουμε για τις συνέπειες που υφίστανται οι γυναίκες σε εποχές κρίσης, συνέπειες που δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά που διορθωτικά ε, ε, έχουν θέση μέσα στον χρόνο και τώρα υπήρχαν ε, ανέκαθεν και τώρα εμφανίζονται με την, με την κρίση. Δεύτερον πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία, είναι απολύτως απαραίτητο. Επιμένω σε αυτή την αναγκαιότητα και τρίτον μου φαίνεται ότι χάρη αυτή την έκθεση θα μπορέσουμε να πράξουμε έτσι ώστε η συμβολή των γυναικών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης να ενισχυθεί περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν άλλη μια φορά να εκφράσω τη στήριξή μου για όλα τα σημεία που υπογραμμίζει η κυρία εισηγητρία από τα στερεότυπα μέχρι την οικογενειακή συνεργασία, μέχρι την ισότητα, τη μισθολογική ισότητα των γυναικών. Ευχαριστώ. Eh, και εγώ προλαβαίνω να πάρω το λόγο λίγο. Έχω ρίξει μια ματιά σε αυτή την έκθεση. Ή, όντως, ε, λίγα σημαντική έκθεση και θεωρώ ότι η οντως ε σημαντικη Μωρίν Σαρτιέ κάνει μια πολύ βασική πρόταση. Δείχνεις πάρα πολύ καλά, ε, φωτίζεις πολύ καλά όλα τα διάφορα στερεότυπα ε, και για τον αγορά εργασίας, τι είναι σημαντικό, τι όχι, το κάνεις πολύ καλά μιλάς για το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα. Επίσης περιγράφεις πώς ακριβώς πλήττονται οι γυναίκες και πώς ε, ε, ε, επηρεάζονται οι γυναίκες από τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες έχουν διαρθρώσει την κοινωνία. Επίσης αναφέρεις τι ακριβώς πρέπει να γίνει και πηγαίνει και αναφέρεις πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αναφέρεις στο σημείο 17 για την συλλογική, ε, για, τις, για τα μαζικά μέσα επικοινωνίας, Φερρυπίν, επίσης για ένα πρόγραμμα δράσης που πρέπει να έχει επιτροπή, επίσης το ότι οι μέλη μειώνουν του προπολογισμού του, πράγμα το οποίο έχει πλήξει Φερρυπίν βαρφονιπιακού σταθμού κτλ. Επίση, υπογραμμίζει τη σημασία για την διαβίου κατάρτιση. Θεωρώ κάνεις μια πολύ σωστή ανάλυση και μια καλή πρόταση που τη συμπληρώνει. Αυτό που μου λείπει και δεν είναι ίσως παράξενο ότι αλήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Εγώ βρίσκω το βασικό πρόβλημα γιατί έχει έτσι η κατάσταση. Ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουμε εδώ στο, στην Επιτροπή. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί έχουμε αυτές, αυτού του είδους πολιτικές. Γιατί έχουμε γραφειοκρατικές οργανώσεις. Έχουμε την Επιτροπή. Ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες που ε, ασκούν κάποια πίεση. Άλλοι αρνούνται. Έχουμε τεχνοκρατική προσέγγιση. Βλέπουμε τα στοιχεία αριθμούς. Μιλάει κανείς για οικονομία ένα μέρος της οικονομίας. Μιλάει κανείς για το δημόσιο χρέος. Η οικονομία όμως δεν είναι δημόσιο χρέος. Η οικονομία είναι όλοι εδώ οι άνθρωποι που βρίσκονται. Ε, ε, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ναι, μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 3%. Αλλά τι, έχουμε 15% ε, ανεργία. Τι κάναμε, αποτύχαμε. Αυτό μου λείπει εμένα. Και για μένα είναι βασικός προβληματισμός. Σίγουρα θα καταθέσω τροπολογίες με αυτή την οπτική γωνία, διότι επαναλαμβάνω, ο βασικός προβληματισμός είναι αυτή που ανέφερα και αυτή οδηγεί στις καταστάσεις που ζούμε. Παρ' όλα αυτά να πω ότι είναι πολύ καλή έκθεση, πολύ σωστή ανάλυση, αλλά λείπει, λείπει, λείπει για μένα αυτό που είπα. Κλείνω εγώ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να πάρει το... Επαναλαμβάνω, η Επιτροπή, μήπως να πάρει το λόγο. Okay. do, you, do you want to floor? No? No? Okay. Όχι. Καλώς. Τότε δίνω το λόγο στην κυρία Μωρίν Σαρτιέ. Ε, παρακαλώ, δικό σας είναι το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που παρενέβησαν την Τζίτα Ε, κυρία Γκρουμάη, σημείωσα αυτό που είπατε, ότι οι γυναίκες μέσω αυτής της κρίσης μπορούν να πάρουν τα ενία, μπορούν να βρουν θέσεις, ε, νέες θέσεις απασχόλησης, ε, σε νέου τύπου θέσεις απασχόλησης, να κινητοποιηθούν ε, στην επιχειρηματικότητα και ειδικότερα όσον αφορά την πράσινη οικονομία αλλά και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όπως βλέπουμε υπάρχουν τομείς που πρόκειται να αναπτυχθούν όπου οι γυναίκες θα πρέπει να βρουν τη θέση τους. Το δεύτερο που σημείωσα είναι ότι επίσης η κρίση έχει γυναικείο πρόσωπο, είναι σιωπηλή αλλά έχει γυναικείο πρόσωπο και ότι πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε ώστε ταυτόχρονα να βγάλουμε τους μεν και τους δε από την κρίση, αλλά ειδικότερα τις γυναίκες. Ευχαριστώ τη Μαρία Γκαμπριέλ για τα όσα είπε. Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα στο οποίο προσπαθώ να οικοδομήσω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για αυτή την έκθεση. Αυτό που ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να επιτύχουμε μια έκθεση η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα όσα λέμε στις διάφορες εκθέσεις. Διότι κάποια στιγμή χρειάζεται να κάνουμε μια συνολική έκθεση των όσων καταγγέλουμε, όλων όσων για τα οποία μαχόμαστε, όλων των θέσεων που μπορούμε να υιοθετήσουμε, ακόμη και αν οι απόψεις, οι ψήφοι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες πάντα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας απαντήσω ότι γνωρίζετε ότι τον αγαπώ πολύ τον πρόεδρό μας της Επιτροπής. Ε, συνεπώς με μεγάλο αίσθημα φιλίας θα του πω όσα πρόκειται να του πω. Ίσως και το γεγονός ότι πλησιάζουν οι γιορτές ε, μου επιτρέπει να πω πράγματα με τρόπο πιο απλό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εγώ σημείωσα με μεγάλη προσοχή την έκθεση προς γνωμοδότηση της κυρίας Τζίμερ που πρέπει να γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε η συγκίτρια για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συμφωνεί με πολλά σημεία που αναφέρονται στη δική μας έκθεση. Η έκθεση της κυρία Ζήμερ ε, επισημαίνει και υπογραμμίζει την καταπολέμηση της φτώχειας, ό,τι πρέπει να κάνουμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό, το πρίσμα υπό το οποίο βλέπει τα πράγματα είναι πιο ευρύ δεν εστιάζεται μόνο στις γυναίκες όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, ε, εστιάζεται ωστόσο και στην ανεπαρκή πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ποιότητας, σε θέσεις εργασίας, απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Εκεί λοιπόν η ανάλυση ε, πλησιάζει και τη δική μας υπογραμμίζει τις περικοπές των δημοσίων προϋπολογισμών Υπάρχει λοιπόν κάποια αντιστοιχεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εγώ θα ήθελα να σας πω είναι ότι είμαι απολύτως διατεθειμένη να προσέξω όλες, να μελετήσω όλες τις τροπολογίες που θα υποβληθούν σε αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσης. Όπως και να έχουν τα πράγματα όλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα μόνο νούμερο. Ότι Τη στιγμή της συνταξιοδότησης, η συνταξιοδότηση των γυναικών είναι 39% χαμηλότερη από αυτή των ανδρών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Ό,τι οδό και αν επιλέγουμε, κύριε Πρόεδρε, αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να μειώσουμε, διότι είναι απολύτως απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα εργαζομένων διαφορετικά. Ευχαριστώ να υπογραμμίσω ότι και εγώ και εγώ και εγώ την αγαπάω την κυρία Μωρίνη Σαρτιέ. Λοιπόν, 9 Ιανουαρίου, 12η ώρα, κατάθεση τροπολογιών. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 18-19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσει η η Επιτροπή μας και για τον Μάρτιο να μπορέσουμε να περάσουμε σε Ολμέλεια. Και θα έχει μεσολαβήσει και 8 Μαρτίου που είναι πραγματικά ε, η πρόταση αυτή θα αποτέλεσει βάση για εκείνον τον εορτασμό, για εκείνη την επέτειο. Ε, εντάξει, συμφωνούμε σε πολλά πράγματα, θα έχουμε όμως και διαφωνίες. Τώρα, αφήνουμε αυτό το σημείο και προς το παρόν διακόπτουμε αφήνω το 12 και πάμε στο 13 γιατί έχουμε ψηφοφορία. Προώθηση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου. Θα δώσω το λόγο σε ποιον. Υπάρχει κάποιος εδώ εισηγητής. Όχι. Άρα, τι. Οπ. Κάτι βλέπω. Τις... Ε, Ποια ήταν η προθεσμία. Όχι, sorry. Amendments. Ε, ε για τις τροπολογίες, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 9 Ιανουαρίου. Okay, we will then start vote. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε unblock. Ξέρω ότι διαφωνούμε σε ορισμένε. Μία-μία θα ψηφιστούν οι τροπολογίες. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Ποια ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία. Τέσσερα. Α. Υπέρ, παρακαλώ σηκώστε τα χέρια κατά, αποχές, εγκρινέται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν. 1,5 λεπτό. <laughs> Κράτησε. Ζητώ συγγνώμη. Okay. Um, we go back to... Uh, Επανερχόμαστε στο σημείο 12. αφορά την προετοιμασία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δίνω το λόγο στην κυρία Γκαμπρίελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη, γιατί εδώ μιλάμε για μια πρόταση γνωμοδότηση. Η επί τη ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, η πρόταση γνωμοδότηση που είχα την τιμή να συντάξω μιλά για τρει ανάγκε. Παρακαλώ, αν θέλετε να συζητήσετε, βγείτε εκτός της αίθουσας. Συνεχίστε παρακαλώ. Συνεχίζω λοιπόν. Τρεις αναγκαιότητες ε, που μας οδήγησαν στη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη εφαρμογής της αρχής ε, οριζόντιου χαρακτήρα όλων των πολιτικών της Ένωσης με τα κράτη εκεί. Δεύτερη ανάγκη η εφαρμογή διατάξεων ρητών υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στις εθνικές νομοθεσίες που θα αποσκοπούσαν αφενός στην εγγύηση του σεβασμού αλλά κυρίως στο να επιτρέψουν την υλοποίηση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών. Τρίτη ανάγκη, η ανάγκη προβολής και επιμένω σε αυτό, προβολής των επιτευγμάτων ορισμένων κρατών ΑΚΕ όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων τη χιλιετία. Ορισμένα κράτη-μέλη πριν από την οριακή ημερομηνία του 2015 έχουν επιτύχει κάποιου στόχου. Πρέπει να διαφημίσουμε τι πρόοδου αυτών των κρατών. Σα υπενθυμίζω ότι μιλάμε για χώρε υποανάπτυξη και δεύτερον να διαφημίσουμε τι βέλτιστε πρακτικέ μεταξύ αυτών των κρατών μαλλών. Βάσει λοιπόν αυτών των τριών αναγκαιοτήτων, οι τροπολογίε μου επικεντρώνονται σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, είναι απαραίτητο να εντείνουμε το gender mainstreaming σε όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ένωσης και κυρίως στη σχέση τη με τα κράτη Α δεύτερον. Μου φαίνεται ότι όλο και περισσότερο η συμπεριλήψη, η συμμετοχή συμβούλων σε θέματα ε, φύλου ή θεματικών υπευθύνων για τι διάφορε πολιτικέ και για τις πολιτικές ασφάλειας και άμυνας είναι απαραίτητο. Τρίτον, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και του υπερασπιστέ των δικαιωμάτων των γυναικών. Και τέταρτον, να προωθήσουμε, να προβάλλουμε το ρόλο κλειδί για τον εκδημοκρατισμό των γυναικών. Το ρόλο κλειδί των γυναικών για τον εκδημοκρατισμό και το ρόλο κυρίω των γυναικών σε όλε τι διαδικασίε επίλυση διενέξεων σε ε, καταστάσεις, ε, σε περίοδους μετά από διενέξεις, μετά από συγκρούσεις. Σε αυτά επικεντρώνονται οι τροπολογίε μου. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων και παραμένω διατεθειμένη ε, να ακούσω τι προτάσει των συναδέλφων που θα μου επιτρέψουν να εμπλουτίσω το κείμενο και θα μου επιτρέψουν να εξασφαλίσω ότι αυτή η γνωμοδότηση τη Επιτροπή για τι Γυναίκε, αυτή την έκθεση τη Επιτροπή Ανάπτυξη θα με βοηθήσει κυρία Γκουρμάη. Θα ήθελα να επιθυμίσω σε όλους ότι για τις χώρες ΑΚΕ είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα στην Επιτροπή γιατί είναι σημαντικό να εντάξουμε την διάσταση του φίλου σε αυτό το θέμα. Και σε σχέση με τη συζήτηση για το πολιτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα είναι κεφαλαίωδους σημασίας για οποιοδήποτε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Επιτροπή ε, ΑΚΕ και με τη συνεισφορά της στην Επιτροπή και με τις εκθέσεις της. Η ε, κυρία Γκαμπριέλ έχει συντάξει μια έκθεση η οποία συνθέτει όλες τις διαφορετικές πτυχές του ζητήματος. Αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει την σημασία της διάστασης του φύλου και της ισότητας των δύο φύλων για την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης είναι σημαντικό που αναφέρεται στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Απλώς θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, πολλές, οι χώρες θα μπορούσαν να κάνουν πολλά, περιπάνω, πολλά περισσότερα από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Αυτή η στόχη είναι το ελάχιστο στο πλαίσιο της ε, ατζέντα για αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θέσει στόχους συναφής με το φύλλο, γιατί οι γυναίκες έχουν κρίσιμη συμμαχησία στην υλοποίηση αυτής της ατζέντα. Είναι σημαντικό που αναφέρεται η επίτευξη του στόχου για την ε, ε, παροχή πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα κορίτσια και στα αγόρια. Είναι σημαντικό να δημοσιοποιηθούν αυτές οι επιτυχίες από την πλευρά της Επιτροπής και είναι επίσης σημαντικό που αναφέρεται στην νομοθεσία τρίτων χωρών, γιατί όταν κάτι θέλουμε να το ε, υλοποιήσουμε στην πραγματικότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και να δημιουργεί μηχανισμούς που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ε, γυναίκες να συμμετέχουν πιο ενεργά στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων. Όχι μόνο στην πολιτική ζωή, αλλά επίση και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκω αυτή την νομοδότηση ιδιαίτερα σημαντική και ευελπιστώ η Επιτροπή ανάπτυξη να την υιοθετήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουρ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την γνωμοδότηση. Να την επικροτήσω. Και θα ήθελα να προσθέσω κάποιες μικρές παρατηρήσεις. Έχω την αίσθηση ότι πιθανώς στην αναπτυξιακή πολιτική θα έπρεπε να έχουμε κάποια πιο εστιασμένη πολιτική. Και όταν λέω πιο εστιασμένη ενώ το ζήτημα της μόρφωσης και της υγείας η εμπειρία που έχουμε από συναντήσεις με τις χώρες και μου λέει ότι έχουμε το θέμα της νησιμότητας των μητέρων συνεπώς η μόρφωση, η εκπαίδευση των μεών, των ε, εργαζομένων ε, σε κοινωτικέ υπηρεσίε υγεία είναι ένα ζήτημα που συνδέεται και η εκπαίδευση αυτή καθεαυτή. Εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι σε πολλέ πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, στα πρώτα σχολικά ε, χρόνια η, εγκατάλειψη, η πρόορη εγκατάλειψη των σχολείων οδηγεί σε χαμηλά μορφωτικά επίπεδα. Συνεπώς αποτελεί ζήτημα κλειδί. Και υπάρχει και ένας άλλος παραγόντας προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε και να βοηθήσουμε σε πολλούς πολλούς τομείς αφήνοντας αυτούς τους ανθρωπιστικούς τομείς ελεύθερους να στην κινέζικη πολιτική. Μου φαίνεται ότι είναι λάθος. Το να έχουμε αυτή την ευκαιρία να διαμορφώσουμε τη μελλοντική πολιτική πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε σε ζητήματα υγείας και μόρφωσης έχοντας υπόψη μας έχοντας υπόψη μας ότι μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο σε αυτούς τους τομείς. Eh, Ευχαριστώ να πω κι εγώ, ε, διότι είμαι στιγιώδης εισηγητής και σε αυτή την γνωμοδότηση. Δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω. Νομίζω η πρόταση είναι καλή. Έχεις κάνει, κάνει και ένα συνδυασμό ε, με τους στόχους που υπάρχουν σε σχέση με το, την ισότητα, ε, την ε, περίθαλψη, τη φροντίδα των μητέρων. Αλλά να πω όμως κάτι ακόμα που θα το προτείνω και δεν θα εκπλαγείς. Υπάρχει και το θέμα για τα δικαιώματα και τη... για τα σεξουαλικά δικαιώματα. Ε, δηλαδή η γυναίκα έχει δικαιώματα η ίδια για το δικό της το σώμα. Να υπογραμμιστεί αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Ε, βλέπω η κυρία εκεί στο βάθος ε, κουνάει το κεφάλι, αλλά Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ε, έχω. Ε, ε, κοιτάξτε, επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να έχουμε απόψεις. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκάμπριελ να ανακεφαλώσει. Ε, Ευχαριστώ τους συναδέλφους, τις συναδέλφισες που μιλήσανε, άκουσα με προσοχή, θα αντιδράσω σε κανένα δύο σημεία τα οποία έχουν όπως αυτό της κυρίας Γκουρμάη για, την ε, βασική, για, την, ε, για το δημοτικό σχολείο, για την εκπαίδευση εκεί. Μου είπε να επιμένω σε αυτό το θέμα, να δούμε για τις χώρες και για αυτό το θέμα, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, η βασική πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπογραμμίζω και όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, είναι σημαντικό να γίνει αυτό Υπάρχουν δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν νομοθεσία στις περισσότερες χώρες, αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας. Ενδεχομένω να έχουν και καλύτερα κείμενα από αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Όμως, όμως αυτά τα κείμενα συστηματικά είναι νεκρό γράμμα. Επίσης δέχομαι με χαρά τις προτάσει τη κυρία Μπάουερ να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση και στην υγεία. Είναι σημαντικά αυτά και Επίσης, δεν χαιρετίζω την πρότασή σας για την σεξουαλική υγεία. Ε, θα δεχτώ με τα χαρά στις ε, προτάσεις σας με τις τροπολογίες. Πρόεδρος, ξέχασα να ρωτήσω αν η Επιτροπή θέλει να, να πάρει το λόγο. Λυπάμαι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, Monsieur Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Προφανώ η Επιτροπή συμφωνεί με την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτέ τι προσπάθειε για τη βελτίωση του φωτικού επίπεδου και τη ε, υγειονομική περίθαλψη για τι γυναίκε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το νομικό πλαίσιο βάσει στο οποίο γίνεται η συνεργασία με αυτέ τι χώρε. Είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και ο, η δικαιολογία, το πλαίσιο είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η συνθήκη τη Λισαβόνα, μετά υπάρχουν η σύμβαση του Κοτονού, η συμφωνία του Κοτονού. Και αργότερα αυτές εξειδικεύονται σε πιο συγκεκριμένα νομικά εργαλεία. Το ζήτημα που θέτει η εισηγήτρια, το ζήτημα τι γίνεται στην πράξη. Όσον αφορά τον γεωγραφικό προγραμματισμό, που αναφέρεται στην έκθεση σε σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Υπάρχουν ήδη συνάδελφοι της Επιτροπής που ασχολούνται με το θέμα και στην προετοιμασία αυτού του προγραμματισμού έχει, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες, προσπάθειες για εκπαίδευση, για κατάρτιση, έτσι ώστε να ενταχθεί καλύτερα το ζήτημα του φύλου στην ε, στην στην εργασία με αυτές τις χώρες. Η νέα οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον επόμενο Μάρτιο, θα προσπαθεί να εντάξει αυτές τις διατάξεις, να, να συμπεριλάβει την υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οριζόντια ζητήματα στην αναπτυξιακή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια και αυτή η υποχρέωση πλέον αναφέρεται και ρητά στην ατζέντα για αλλαγή, που είναι και το πλέον πρόσφατο έγγραφο ε, πολιτικής που μας καθοδηγεί στο ζήτημα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης, επίσης να υπογραμμίσω κάτι που αναφέρεται και στις συμφωνίες του Κοτονού υπάρχει μια αναφορά στο ζήτημα του, του φύλου, της διάστασης του φύλου στην ανθρωπιστική δράση. Καθώς. Γιατί επίθετο και το ζήτημα της μετάβασης από την ανθρωπιστική δράση στην αναπτυξιακή συνεργασία. θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμών και ειδικών πάνω στα ζητήματα του φύλου στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ και στον προϋπολογισμό. Το προϋπολογισμός προτείνει επιτροπή είναι 34 ε, δισεκατομμύρια. Γνωρίζετε ότι αυτές οι δημοσιονομικές αυτά τα δημοσιονομικά ζητήματα ρυθμίζονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο να παίξει για να υποστηρίξει αυτή τη θέση της Επιτροπής. Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω το εξή. Στην πρόταση τη Επιτροπή, όπω ήδη το γνωρίζετε, προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν αξιολογήσει, εμπειρογνώμονε, αναλυτικέ εκθέσει, να υπάρχει παρακολούθηση τη εξέλιξη. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι στα χέρια τη Επιτροπής. Και γνωρίζετε ότι σήμερα, όπω έχουν τα πράγματα, το 2% προσφε... Ε, τα κράτη-μέλη το 2, προσφέρουν το 2% για αναπτυξιακή συνεργασία, κάτι που είναι λίγο. Δεν επαρκεί. Το βλέπουμε στη συνεργασία με τις ε, χώρες και το επίπεδο που χρηματοδότησης που παρέρχεται παρέχεται στην Επιτροπή είναι χαμηλό και η Επιτροπή προτείνει να ανέλθει στο 5%. Η εισηγήτρια στην Επιτροπή ΤΕΒΕ Ανάπτυξης έχει συμφωνήσει με το θέμα αυτό και ευελπιστώ ότι θα τη συμπεριλάβει στην γνωμοδότησή τη. Βρισκόμαστε στη θέση σα για να σα δώσουμε περισσότερε πληροφορίε. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να πω για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την κατάσταση πολεμιών 9 Ιανουαρίου 12. 21 Ιανουαρίου ψηφίζουμε και η Επιτροπή Επανάπτυξη ψηφίζει στις 19 και μετά περνάμε στην Ομέλεια. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο για τη μερικέ διατάξει είναι η κατάσταση των γυναικών στη Βορεια Αφρική. Στη Αφρική. Το... Θα μιλήσει η κυρία Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχαριστήσω για τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή για τις γυναίκες. Είτε με το Λίρινγκ όπως κάναμε στην αρχή, συμμετείχαν σημαντικές γυναίκες και στη συνέχεια η δική μας ε, αντιπροσωπεία στην Τινησία και ο Πρόεδρος Γκούσταυσον και οι συναδελφοί Γκαμπρίελ και Νίλσεν ήταν εκεί και πιστεύω ότι, ότι με αυτή την άμεση επαφή καταλάβαμε πολλά ακούγοντα άμεσα τη φωνή των γυναικών. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να συλλεξώ και άλλα πολλά στοιχεία άμεσα και έμεσα από ενδιαφερόμενους, από σημαντικές γυναίκες ε, και κυκλοφορήσαμε και ένα ερωτηματολόγιο μεταξύ σημαντικών γυναικών σε διάφορες χώρες συγκεκριμένο και η έκθεσή μου ουσιαστικά επικεντρώνεται σε τέσσερις χώρες για τις οποίες μιλήσαμε. Τις τέσσερις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Αίγυπτος, την Λιβύη και Μαρόκο. Η σημερινή μέρα είναι σημαντική, διότι ακριβώς πριν από δύο χρόνια, στις 18 Δεκεμβρίου, ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στην Τινησία που οδήγησαν στα μεγάλα κινήματα, επαναστατικά θα λέγαμε, με τη συμμετοχή πολυάριθμων γυναικών νέων της επωνομαζόμενης ε, ε, Αραβικής Άνοιξης. Θα θυμάστε στις 17 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν όλα αυτά στη Δινησία πριν από δύο χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιν μιας ιδιαίτερα σύνθετης κατάστασης, ε, διαρκώς μεταλλασσόμενης, Παρότι η εκθέση μα ε, μας έγινε πριν από ένα μήνα και η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς. Είναι εντελώς ρευστή και δυστυχώς ε, διαβλέπουμε ανησυχητικές ενδείξεις. Αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή θεσμική και πολιτική κρίση στην Αίγυπτο με ε, την προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών από τον πρόεδρο Μόρση, ο οποίος είχε συμβάλει στη διαμεσολάβηση στη Γάζα και τώρα θέτει σε δημοψήφισμα ένα σχέδιο συντάγματος στην Αίγυπτο που έχει το ελάττωμα ότι είναι σχέδιο της πλειοψηφία. και σε αυτή τη μεταβατική στιγμή, τη δύσκολη μεταβατική στιγμή η διαδικασία που λαμβάνει η χώρα σε όλες τις χώρες εκτός από το παρόκο που το έχει ήδη εγκρίνει θεωρεί ότι ε, θα πρέπει να, είναι ένα σχέδιο στο οποίο να συμμετέχουν όλοι οι πληθυσμοί. Αυτό πρέπει να συμβεί και στην Τινησία και στη Λιβύη. Να έχει τη συμμετοχή όλων των πληθυσμών. Η απειλή είναι ότι και στην Τινησία έγιναν σημαντικά γεγονότα. Τον Αύγουστο είχαμε μια επανάσταση σε πλατείες με συμμετοχή πολλών γυναικών και μη κυβερνητικών οργανισμών όσον αφορά τον κίνδυνο τροποποίησης του άρθρου 1 αυτό το θέμα εκρεμεί ακόμα στην Τινησία. Αφορά την βούληση του κόμματος της πλειοψηφίας, του ΕΝΑΝΤΑ, να εισαγάγει τη Σαρία όχι ως ε, την αναφορά στην ε, Ισλαμική θρησκεία, όχι ως θρησκεία της πλειοψηφίας του πληθυσμού, αλλά ως νομοθετικής βάσης. Σε αυτό παίζονται πολλά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες και την κατάστασή τους. Γνωρίζουμε πράγματι ότι υπάρχει κίνδυνος επανάστασης όσον αφορά τον ίδιο τον ορισμό του νομικού καθεστώτος, των δικαιωμάτων και της ισότητας ως θεμελιδών αρχών που αφορούν την κατάσταση των γυναικών στο πλαίσιο οικουμενικών δικαιωμάτων όπως το έχει ζητήσει η κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο και στην Τινησία. Ε, Ρητά. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αντιμετωπίζοντας αυτές τις πραγματικότητες. Εγώ θα ήθελα να είμαι ελάχιστα διπλωματικά. διπλωματική. Πρέπει να αποφύγουμε το σφάλμα που έγινε και από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εντός του πολιτικού Ισλάμ υπάρχουν διάφορα ρεύματα. Δεν υπάρχει μόνο ένα Ισλάμ. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν διάφορα ρεύματα, μετριοπαθείς, συντηρητικοί και άλλοι προσπαθούν να παρέχουν εκχωρήσεις σε σαλαφιστές, ριζοσπαστικούς, όλα αυτά γίνονται στην Δυνησία κυρίως και στην Αίγυπτο. Ξέρουμε ότι το βλέμμα της Ευρώπης πρέπει να γίνει πιο ευρύ πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο και το έχω συμπεριλάβει στην εκθεσή μου την αιρεσιμότητα όσον αφορά τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα, το, την αρχή more for more σε εταιρικέ σχέσεις, σε συνεργασία. Δηλαδή υποστηρίζω το να προσέξουμε και να σεβόμαστε την ε, συμμετοχή, την ε, χειραφέτηση των γυναικών. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πιο ευρύ βλέμμα διότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι χώρες περιορίζονται έντονα από τα φονταμεταλιστικά του στοιχεία, την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και από το Κοτοάρ για τους αδερφούς μουσουλμάνους και θεωρώ ότι και προς αυτές τις χώρες η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει μια δράση. Όπως βλέπετε αυτό το ενσωματώνω κατά κάποιο τρόπο στην εκθεσή μου διότι είναι αποκύημα των προβληματισμών που ακολούθησαν τα τελευταία γεγονότα τα οποία μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε ένα μεταβαλλόμενο σενάριο. Όσον αφορά το ζήτημα της εκθέσης, εγώ προσπάθησα να αναδείξω τέσσερις σημαντικούς στόχους. Όσον αφορά την κατάσταση της γυναίκας, πρώτα απ' όλα ποια είναι η πρόοδοι, αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι όσον αφορά την κατάσταση της γυναίκας σε αυτές τις τέσσερις χώρες, ποιο είναι το επίπεδο χειραφέτησης των γυναικών, συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών, στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, στα μέσα μαζική ενημέρωση που έχουν στρατηγικό ρόλο να παίξουν σε αυτή τη δημοκρατική μετάβαση, τι δυσκολίε και τη πιθανά εμπόδια, όπως ξαναείπα, που έχουν αυξηθεί δυστυχώ και ποια μέσα πρέπει να υλοποιήσει, να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των γυναικών και την ισότητα των φύλων στη δημοκρατική διαδικασία. Για να σας το πω συνοπτικά, εμείς βρισκόμαστε ενώπιον επίσης ενός κόμβου όπου θα μπορούσαν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι γυναίκες. Ε, έχουμε και ένα προβληματισμό που αναπτύσσεται μεταξύ γυναικών του Ισλάμ. Αυτή η προσπάθεια να αναγνώσουν αυτόνομα τις σχέσεις μεταξύ Ισλάμ και δημοκρατίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πιο ανοιχτό μυαλά αυτό του είδους η σχέση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία στην οποία μπλέκονται διαφορετικά οι γυναίκες στην Τινησία παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνταγματική διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Οι γυναίκες ε, στην Αίγυπτο βρίσκονται στο περιθώριο, στο Μαρόκο υπάρχει κάποια συνένεση από τις γυναίκες και στη Λιβύη που είναι μια ζώνη που μέχρι στιγμής ε, παραμένει σκοτεινή και εγώ είχα τη χαρά να γνωρίσω βουλευτές της Λιβύης ε, και αυτή τη στιγμή και Γενική στο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, το μη θρησκευτικό κόμμα και υπάρχουν γυναίκε στο κοινοβούλιο, ενώ παλιά ήταν αποκλεισμένε εντελώ. Υπάρχουν δηλαδή φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Τώρα, στα συντάγματα το ισχυρότερο αίτημα είναι για δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεγάλη συζήτηση αφορά την αναγνώριση των διεθνών συνθήκων και η συγκεκριμένη εφαρμογή τους, όπως είπε για τις χώρες και προηγουμένως η, η κυρία Γκαμπριέλ. Υπάρχουν πολλοί νόμοι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όμως. Και αν δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης και ελέγχου, παραμένουν νεκρογράμμα αυτά τα συντάγματα. Ένα κομμάτι παλιάς ρητορική. Θεωρώ ότι το θέμα λοιπόν εδώ είναι να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία χειραφέτησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Ένα μεγάλο ερώτημα, σημαντικό, είναι να δούμε πώς οι γυναίκες συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε κοινωνικό επίπεδο και την κοινωνική τους χειραφέτηση. Και εδώ είναι ενδιαφέρον αυτό το πλαίσιο, το σκοτεινό και φωτεινό πλαίσιο, αυτές τις σκοτεινές και φωτεινές πτυχές. Στη Λιβύη, για παράδειγμα, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι γυναίκες στα πανεπιστήμια είναι περισσότερες από τους άντρες, όπως και στην Τινησία, ενώ στο Μαρόκο είναι πολύ λιγότερες όσον αφορά την γυναικεία παιδεία, μόρφωση. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικέ ταχύτητε και διαφορετικά μέσα. Η οικονομική αυτονομία. Εμεί έχουμε πραγματικότητε, ε, ε, παραδείγματα επιχειρηματικότητα ε, και μικρή ακόμα, ειδικότερα στην Τινησία, στη Γεωργία για παράδειγμα, αλλά και στην Αίγυπτο. Την αίσθηση ότι εδώ έχουμε οπισθοχωρήσει λόγω τη οικονομική κρίση και ο περιορισμό των πιστώσεων. Υπό αυτή την έννοια οι μικροπιστώσει, μια εμπειρία πολύ ενδιαφέρουσα στην Τινησία, όπου συμμετείχαν ήδη 2.000 γυναίκες με ενώσεις βασικές ε, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Για παράδειγμα, προτείνοντα την Παγκόσμια Τράπεζα να υποστηρίξει ε, εγκυτικά κονδυλέ για τις τι ε, χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστεί με τα μέσα που έχει, αλλά να τα χρησιμοποιεί όπως είπε προηγουμένως η Κομισιόν, ότι στο εσωτερικό του μεγάλου προγράμματος ανα, ανάπτυξης ε, και προπολογισμού του 2014-2020 θα μπορούσαν να υπάρχουν πόροι ώστε οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά μέσα ανάλυσης, παρέμβασης και ειδικών εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα ζητήματα. Η μάχη σε αυτές τις χώρες θα νικηθεί σε μεγάλο βαθμό σε περιφερειακό και εδαφικό επίπεδο. Η ιδέα ότι όλα θα επιληθούν στις μεγάλες πόλεις σε εθνικό επίπεδο ενέχει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης ε, των ικανοτήτων ότι θα είχαμε τις ικανότητες να λύσουμε πράγματα σε σχέση με τις εδαφικές δυνατότητες. Δεν πρέπει να υπε... παραμελούμε το ζήτημα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας διότι υπάρχει ελάχιστη δικαιοσύνη για αυτές τις γυναίκες και υπονομεύεται η ασφάλεια όλο και περισσότερο. Δυστυχώς κάθε μέρα στυλιτεύονται για τον τρόπο που ντύνονται, για ειδικά από τους φονταμενταλιστές και κοινωνικός διαχωρισμός, για παράδειγμα σχολεία αγοριών κοριτσιών. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τις γυναίκες ε, της γενιάς μεταξύ 40 και μεγαλύτερων ως οπισθοχώρηση, αδιανόητη. Μας το είπαν πολλές γυναίκες θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τι συνθήκε ελευθερία. Πιστεύω επίση ότι το άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι εκείνο τη σωστή συνεργασία τη Κομισιόν στο πλαίσιο των εκθέσεων με το UN Women των Ηνωμένων Εθνών που έχει δημιουργήσει έδρες, έχει δημιουργήσει αντιπροσωπείες και στις τέσσερις χώρες εκτός από τη Λιβύη, όπου πρόκειται τώρα να ε, εγκαθιδρυθεί και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το πιέσουμε να γίνει, διότι εμπλέκονται δίκτυα ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε ως δέσμευση μεταξύ όλων των δεσμεύσεων στη διμερή συνεργασία το θέμα του more for more όσον αφορά τα δικαιώματα και την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών πρέπει να είναι απολύτως παρόν σε κάθε διμερές πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι από το 2012 η Κομισιόν υποστήριξε με 91 δισεκατομμύρια ευρώ τη συμφωνία με την ε, UN Women και το περιφερειακό πρόγραμμα που ονομάζεται Spring Forward for Women που θέλει να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους ε, για τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Και τα η δική μας μέθοδος εκδημοκρατισμού μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό σημείο μαζί με το νέο Ταμείο Υποστηρίξης της Δημοκρατίας. Εγώ πρότεινα και εδώ κλείνω ότι συμβολικά αλλά όχι μόνο αξίζει να παρακολουθούμε την κατάσταση των γυναικών κάθε χρόνο το Μάρτιο καλό θα ήταν να αφιερώνουμε μία συνεδρίαση για την κατάσταση των γυναικών στην ε, συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πολύ θετικά βλέπω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΒΕ που υπενθυμίζει κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά πραγματικά πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψει κανείς με λίγα λόγια. Ξέρετε ότι 6.000 ε, λέξεις ήταν ε, το όριο. Εγώ είμαι στη διαθεσή σας για σχόλια Ευχαριστώ. και θα μπορούσα να τα ενσωματώσω να τα συμπεριλάβω στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την Επιτροπή μας για την πρωτοβουλία αυτή της σύνταξης έκθεσης και την εισηγήτρια φυσικά την κυρία Κώστα η οποία έχει πολύ εμβαθύνει στο θέμα και το αντιμετωπίζει με μεγάλη δέσμευση όπως φάνηκε από την παρουσίασή της. Θεωρώ πολύ σημαντικό να συγκρατήσουμε κάποια σημεία. Πρώτον ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, αναφέρθηκε σε αυτό η συγγήτρια Υπάρχουν χώρες στις οποίες υπήρχε μια υποδομή δικαιωμάτων των γυναικών, όπως είναι η Τινησία, και υπάρχουν και χώρες όπου η παράδοση, η, ο ε, ε βάρεναν περισσότερο όπως είναι η Αίγυπτος, η περίπτωση της Αιγύπτου. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ε, καταγράφει η ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια παντού. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε έστω στην Αραβική Άνοιξη που ήταν μια έκφραση κοινών στόχων, κοινών αξιών από τους αραβικούς λαούς. Ξεκινάμε με άλλη αφετηρία για το ρόλο και τη θέση που έχουν οι γυναίκες σήμερα. Το άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι γυναίκες στην ε, Αραβική Άνοιξη οι οποίες έκαναν τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ήταν μια μικρή μειοψηφία. Στις περισσότερες χώρες και οι περισσότερες γυναίκες κάναν τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία. Κάναν τον αγώνα για δικαιοσύνη, για συνθήκες αξιοπρέπειας ε, στην αγορά εργασίας, για, για την ανάγκη ελευθερίας στο να, στο ασκούν τη, τη θρησκεία τους, το Ισλάμ Γι' αυτό πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, πώς προσεγγίζονται και είναι πολύ σημαντικό και οι μελέτες που έχουν γίνει σήμερα και οι, αναφορέ αναφορές από μελετητές εννοώ στις ίδιες τις χώρες που ζουν την πραγματικότητα, γιατί καμιά φορά εμείς τα βλέπουμε λίγο ομοιόμορφα και ισοπεδωμένα από τη δική μας σκοπιά. Άρα υπάρχει σε αυτέ τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν σήμερα, όπου χτίζεται κάτι καινούριο, με τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες χώρες, να ενθαρρύνουμε και το διάλογο για τα γυναικεία θέματα, για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί δεν είναι παντού παρόν ο διάλογος. Στην Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη, δεν βγαίνουν στην πλατεία χρήρ οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, βγαίνουν να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Σαρία. Λοιπόν, χρειάζεται μια προσέγγιση και επιστημονική και ε, κατά περίπτωση σε αυτή την, ε, σε αυτή την ε, προσπάθεια που, που εμείς κάνουμε να ανοίξουμε τις ευκαιρίες της γυναίκες για αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία που ανέφερε η συγκήτρια. Ο ΙΕ, είμαστε πέρυσι κύριε Πρόεδρε και θυμόσαστε και στην Ουάσινγκτον μαζί με την τελεγκασιόν της Επιτροπής μας και έχουν και αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί την ανάγκη να συνεργαστούμε για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Κυρία Μπατσλέ, όταν μας επισκέφθηκε στην Επιτροπή μας, μας είπε ότι φεύγει για την Αίγυπτο την επομένη, ακριβώς για αυτά τα θέματα. Έχουμε συνομιλητές, έχουμε εργαλεία σε διεθνές επίπεδο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Η World Bank και όλα αυτά. Από την άλλη μεριά η Ευρωμεσογειακή Συνέλευση η συνέλευση αυτή, η Επιτροπή Γυναικών, στην οποία συνέβαλα και εγώ, αν μου επιτρέπετε, στη δημιουργία αυτής της Επιτροπής, ήταν μια πολύ θετική έκπληξη για μένα. Φυσικά δημιουργήθηκε πρώτη Αραβικής Άνοιξης και σήμερα θα έλεγα επειδή τα κοινοβούλια από τις χώρες Αραβικής Άνοιξης δεν είναι καλοί συνομιλητές μας διότι βρίσκονται σε συντακτική αναθεώρηση, δεν λειτουργούν ε, κανονικά αλλά και στην προηγούμενη κατάσταση ε, στα προηγούμενα καθεστώτα όταν άρχισε η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα κοινοβούλια των χωρών από την απέναντι όχθη υπήρχαν γυναίκες αποφασισμένες για την αλλαγή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των γυναικών, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για την πρόσβαση στην παιδεία. Και σήμερα εκπλήσωμαι όταν βλέπω γυναίκες στο Μαρόκο να κάνουν εισηγήσει και να δίνουν αγώνα για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Τον αγώνα δηλαδή που δίνουμε και εμείς στο Βορρά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν και πολλά πεδία συνεργασίας, διότι ενθαρρύνονται από την δική μας συνεργασία, ανταλλάσσονται καλές πρακτικές και χρειάζεται πια να, κάνουμε μια, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια αξιολόγηση όλων των πόρων μέσα από την πολιτική γειτονία που πηγαίνουν στις χώρες αυτές, το SPRING, το νέο ε, χρηματοδοτικό εργαλείο και επίσης ε, ε, όλα τα άλλα εργαλεία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Επίσης, ο νέος ο, ε, εκπρόσωπος της κυρίας Άστον, ο κύριος Λαμπρινίδης, πρέπει, νομίζω δεν θα έχει αντίρρηση ο ίδιος, πρέπει και αυτός να εντάξει στις προτεραιότητές του την ε, θέση των γυναικών όταν παρακολουθεί, καταγράφει, ενημερώνει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται, θέλω να πω, μια κινητοποίηση αλλά από όλους τους διεθνείς φορείς ε, και με όλα τα εργαλεία που έχουμε και να μην ξεχάσουμε επίσης ε, όταν θα ολοκληρωθεί η έκθεση μπορεί να έχουμε και εξελίξει στη Συρία να εντάξουμε στην προβληματική μας και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και την Ιορδανία που βρίσκεται σε αναβρασμό η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν θα παρέμβουμε στην εξέλιξη της ε, κοινωνικής ε, αυτής αναταραχής, αλλά θα μπορούμε να πούμε ότι στηρίζουμε παντού τον αγώνα που δίνουν οι γυναίκες για την αξιοπρέπεια, την δημοκρατία, την ευημερία και τα δικαιώματά τους διότι η ιστορική εμπειρία μας λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχημένη μετάβαση, επιτυχημένη μετεξέλιξη πολιτική και κοινωνική, αν δεν στηρίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και δεν αξιοποιεί σε αυτή την μετεξέλιξη της κοινωνίας το ανθρώπινο δυναμικό που είναι οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ. λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα απόλυτα με την κυρία Ισηγήτρια. Πρέπει να προσέχουμε εμείς στην Ευρώπη όταν μιλάμε για αυτούς τους τόπους. Διαφέρουν μεταξύ τους συνταγματικά και οι προσεγγίσεις τους είναι διαφορετικές με τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, η Αραβική Άνοιξη και οι ελπίδες που μας προκάλεσε τότε και το μέρο όπου βρισκόμαστε σήμερα, κατανοούμε προς τα που οδεύουν. Έχουμε ανοίξει ένα τρομακτικό κουτί της Πανδώρας τώρα, ειδικότερα για τις γυναίκες. Αναφέρατε όλοι για την Αίγυπτο και εγώ γνωρίζω από εμπειρία μου ότι είναι μια χώρα που θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών ουσιαστικά όπως τον δρομούν. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην Αραβική Άνοιξη σήμερα είναι τρομοκρατημένες, θα θυματοποιηθούν και το θετικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τις προστατεύσουμε θα ήταν να τονίσουμε την ευαισθητοποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο για το ποιες είναι αυτές οι γυναίκες ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να θυματοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπους προστασίας τους μέσω των δικών μας συζητήσεων εδώ. Ένας πρακτικός τρόπος θα ήταν αν είχαμε προσωπικά χρήματα και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χρήματα ο καθένας μας για να διεξάγουμε μια μικρή σύνοδο εκεί, αν μπορούμε να έχουμε το θάρρος να το κάνουμε. Με αυτές τις γυναίκες, ας τις αναδείξουμε, ας τις ε, προβάλλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήταν πολύ χειρό αυτό. Ένα από τα πράγματα που δεν αναφέρεται είναι τα ζητήματα των ομοφιλοφίλων των LGBT. Τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τις ε, λεσβίες γυναίκες. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ έκανα μια ομιλία στην Ουγκάντα όπου τώρα τον ε, είναι μια γυναίκα λεσβία τιμωρείται με διαβίω φυλάκιση, με ε, ισόβια κάθριξη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις ενισχύσεις, τις βοηθείες, τη πακέτα Θα πρέπει να φροντίζουμε να καταλήγουν στους σωστούς αποδέκτες, να χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτά είχα. Νομίζω να πω. Θα πρέπει να με συγχωρέσετε γιατί πρέπει να αναχωρήσω, αλλά σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους. Μετά από αυτές τις θλιβερές, δυστυχώς, ειδήσει. Καλά Χριστούγεννα και σε εσά. Έχουμε πολλούς στην, ε, στον κατάλογο μιλητών. Τέσσερα άτομα. Και θέλω να δώσω το λόγο και στην Επιτροπή. Συνολικά έξι θα μιλήσουν. Έχουμε 17 λεπτά στη διάθεσή μας πριν να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Θα σας ζητήσω λοιπόν να είσαστε έτσι σύντομοι για να μπορέσουμε να τελειώσουμε ε, ε, στην ώρα μας και να μην ξεπεράσουμε και το χρονοδιάγραμμα για τους ε, Η κυρία Κιλ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τη συνάδελφό μας για το έργο της που όσον αφορά την, την Ισία αντικατοπίζει πολύ σωστά τις ανταλλαγές που είχαμε στις αντιπροσωπείες των γυναικών όταν πήγαμε εκεί στη χώρα. Δύο σημεία στα οποία προβληματίζουμε θα ήθελα δεν να σας πω μήπως θα ήταν κατάλληλη στιγμή ήδη επροτάθη από μία συνάδελφο για τα δικαιώματα των φιλοφίλων εγώ θέλω να προτείνω μια τροπολογία ε, έχει να κάνει με τη για τον ακροτηριασμό των γυναικείων οργάνων κάτι που γίνεται σε αυτές τις χώρες το βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία και με το ε, σώμα των ιατρών. Θα πρέπει να δούμε, είναι κάτι το οποίο συζητάμε πολύ συχνά για την υποσαχάρια Αφρική. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ε, βασικά αυτά όλα ξεκινάνε από την Αίγυπτο. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω μια τροπολογία πάνω σε αυτό το θέμα, ακροτηρισμό γεννητικών οργάνων δηλαδή, αν συμφωνείτε κι εσείς. Ευχαριστώ. Επόμενος στη λίστα η κυρία Νικολάη. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου του ΑΛΔΕ, διότι εγώ είμαι σκιώδη για αυτή την εκθέση. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Κώστα για αυτή την εκθέση. Είναι πολύ ισορροπημένη και αγγίζει πολλά σημαντικά ζητήματα όπως τη συμπεριλήψη της ισότητας των φίλων στο Σύνταγμα ακόμη και στο προηγούμενο Σύνταγμα ήταν καλύτερη η ισότητα των φύλων. πολέμηση της ατιμορρησίας σε περίπτωση διαφορών φύλων κτλ. Ε, θα ήθελα να τονίσω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζαν οι γυναίκες στην Αραβική Άνοιξη. Δυστυχώς ε, στην αρχή ξεκίνησαν αυτό τον τρόπο επανάστασης οι γυναίκες και μετά κινδύνεψαν να χάσουν να είναι χαμένη των αλλαγών. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι η, σημα... η σπουδαιότητα της θρησκείας. Αυτή η αραβική άνοιξη έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα συμβατότητας μεταξύ δημοκρατίας και κοσμικής κοινωνίας. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πραγματική δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα σε μια χώρα όπου αρχίζει αρχίζει να αναπτερώνεται η κοσμική κοινωνία. Είδαμε τι έγινε στην Τινησία, είδαμε τι έγινε στην Λιβύη, στην Αίγυπτο. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε να έχουμε μια εκστρατεία εγκύρης ευαισθητοποίησης ώστε να ξεκινήσουμε ξανά να μαχόμαστε υπέρ του ρόλου των γυναικών διότι πολλές ενδείξεις υπάρχουν ότι υπάρχει μια τάση αποφυγής του σεβασμού του ρόλου των γυναικών. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα επιπλέον σημείο σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία, στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Αλλά η Συρία είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο. Ίσως θα μπορούσαμε όλοι μαζί να κάνουμε κάποια δήλωση πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μιλήσουμε για τις γυναίκες της Συρίας και ίσως να κάνουμε έκκληση ειδικά σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη περίοδο διότι κάθε μέρα στις ειδήσει βλέπουμε να πεθαίνουν γυναίκες και παιδιά σε αυτό το εμφύλιο πόλεμο θα ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν μπορεί να ευαισθητοποιήσει κόσμο Έχω κάποιες τροπολογίες, αλλά σε γενικές γραμμές ε, η έκθεση είναι πολύ καλή και ε, εγώ επικροτώ το να μελετάμε αυτή την κατάσταση των γυναικών στην Αφρική, στη Βόρεια που για μας τους φιλελεύθερους και, αλλά και για όλους μας ουσιαστικά ε, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία Ζάμποσκα. Παρακαλώ. Uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έχουν πολλά λεχθεί από αυτά που ήθελα εγώ να αναφέρω. Επομένω θα περιοριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Κώστα για την έκθεση που προετοίμασε. Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη η έκθεσή της. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το ζήτημα που προσπαθεί να πραγματευτεί σε αυτή την έκθεση και ε, ε, ε αναφέρεται σε ζητήματα τα οποία είναι και πολλαπλά, αλλά επίσης και ε, είναι χρόνια και από τις, τα συνήθεια στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα ασταθής. Μια περιοχή στην οποία η περιφερειακή κατάσταση αλλάζει καθημερινά. Όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο. Βλέπουμε ότι και σε σχέση με το καθεστώς των γυναικών υπάρχουν πολλά κύματα αλλαγής μερικές φορές προς το καλύτερο, μερικές φορές προς το χειρότερο. Τη δεκαετία του 80 εργαζόμουν στο Αλγέρι και έμεινα εκεί τέσσερα χρόνια. Είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω πολλές πτυχές της κατάστασης των γυναικών εκεί. Σε πολλές πτυχές μάλιστα η κατάσταση των γυναικών εκεί ήταν καλύτερη από σήμερα. Και το οποίο τελικά έχει σχέση με το ποιο βρίσκεται στην εξουσία, ποιο ελέγχει τι κοινωνικέ δομέ κτλ. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν θέτουμε ποια είναι τα αιτήματά μας, ποιες είναι οι απαιτήσει μας από αυτή την περιοχή. Πρέπει. πρώτα απ' όλα να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπιών, πολιτιστική αλλαγή. Όταν μιλάμε για ζητήματα όπως η εμπορία ανθρώπων ή ο ακροτηριασμός γυναικείων γενετικών οργάνων ή η ο ακροτηριασμος γενικων γενετικων οργανων κατά των γυναικών, είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα και πρέπει να τα θέτουμε και πρέπει να τα καταδικάζουμε, αλλά επίση υπάρχουν και θετικέ πτυχέ τι οποίε πρέπει να αναδείξουμε σε αυτέ τι κοινωνίε. Είχα την ευκαιρία, για παράδειγμα, να διαπιστώσω ότι είναι ιδιαίτερα ισχυρή η οικογενειακή δεσμή, η πυρηνική οικογένεια. Έχει σημαντικό ρόλο και βοηθά τις γυναίκες ε, ενίοτε να ξεπερνούν σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό που λέω είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη καθώ επίση και οποιαδήποτε προσπάθεια υποστήριξης ε, είναι ε, ιδιαίτερα περίπλοκη. Μερικέ φορέ η προσέγγιση μα μου φαίνεται υπερβολικά ιδεαλιστική, ίσω να του ζητάμε υπερβολικά πολλά. Γιατί εμεί είχαμε τη χαρά επί δεκαετίε να ζούμε σε μια ειρηνική ήπειρο, να απολαύσουμε του καρπού τη δημοκρατία γιατί που δεν ισχύει για εκείνε τι περιοχέ. Θα προτείνω τροπολογίε. Ευχαριστώ. Καλώς ο μιλητή να πάρει το λόγο η Επιτροπή είμαι εγώ, είμαι σκιώδη ο και σε αυτή την έκθεση όπως όλοι οι άλλοι συγχαίρω την συγγήτρια για μια πολύ καλή έκθεση έκανε συλλικνά πολύ καλό έργο, μια σωστή ανάλυση έχει συμπεριλάβει πολλά πράγματα όπως είπε, είναι περίπλοκο το θέμα δεν είναι και τόσο εύκολο Καλύπτει πολλού τομεί που είναι σημαντικοί για τις θέσεις μας και υπάρχουν μια σειρά πραγμάτων που είναι καλά. Το δίνεις βάρος στην ε, νομοθεσία για τα δικαιώματα των γυναικών. Ότι στην νομοθεσία θα πρέπει να δει κανείς και το θέμα της σεξουαλικής βίας εις βάρος των γυναικών. Επίσης διασαφηνίσει θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, περίθαλψη της ε, μητέρες και όταν μπαίνει σε τομείς που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή γυτνίαση και τις δράσεις της Ευρώπης ε, λες ότι εμείς στη σχέση μας με αυτές τις χώρες θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας για την εξωτερική πολιτική. Πάρα πολλά είναι τα θετικά να πω όμως δύο σημεία στα οποία εγώ σίγουρα θα καταθέσω τροπολογίες. Όταν λέμε για, τη για τον εκδημοκρατισμό, για αυτή τη διαδικασία. Άλλοι μπορεί ή και ίδιοι ακόμα μπορεί να μην θεωρούν ότι είναι εκδημοκρατισμός αυτό που γίνεται, ότι είναι μια διαδικασία πολιτική. Αναρωτιέται όμως κανείς, είναι εκδημοκρατισμός όταν δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να συμμετέχουν. Για μένα είναι όχι η απάντηση. Αναγνωρίζω ότι είναι μια δράση, μια εξέλιξη πολιτικής φύσεως. Δεν ξέρω, θα δούμε για άλλους μήπως μπορούμε να εκφραστούμε πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο στο G για την πολιτική γυτνίαση, όπου πρέπει να δοθεί έμφαση για την ισότητα ανθρώπων γυναικών. Εγώ θα έλεγα όχι μεγαλύτερο βάρος. Θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι θα είναι σημείο εκκίνησης. Έχουμε να κάνουμε το άρθρο 8 της συνθήκης της Τσαβάνος ότι όλα τα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βάλουν υπόψη αυτό. Όχι ότι λέμε ότι επιθυμητό κτλ. Ότι είναι βασικό αίτημα. Τέλος πάντων, να συγχαρώ για μια πολύ καλή εργασία και προσδοκώ στη συνέχεια αυτού του έργου και τώρα με μέγιστο 1,5 ε, λεπτό οι επόμενοι δύο ομιλητές. Α, συγγνώμη, ξέχασα την κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πάρω το λόγο οπωσδήποτε διότι είχα πάει στην Τινησία με την κυρία Συγήτρια και χαίρομαι που βλέπω ότι οι ανταλλαγέ που είχαμε εκεί αντικατοπτρίζονται στο κείμενό τη. Δύο σημαντικά πράγματα υπάρχουν στο κείμενό τη. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύει ορισμένα κεκτημένα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στι ε, σχετικέ χώρε. Αφετέρου, κυρίω το κείμενό τη μα επιτρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για κάποια θέματα. Τέσσερα σημεία. Ναι στη συμμετοχή των γυναικών στη μεταβατική διαδικασία, αλλά έκκληση για την ανάγκη χρηματοδότησης εκπαιδεύσεων, καταρτήσεων για να προετοιμαστούν οι γυναίκε για την πολιτική ηγεσία και κυρίως να βγούμε από τις πρωτεύουσε αυτών των χωρών να πάμε στις περιφέρειες ώστε να δούμε γιατί επανέρχονται τα Ισλαμιστικά κόμματα στην εξουσία. Δεύτερον, προγράμματα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, να ενεργοποιηθούμε και εκεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τρίτο σημείο, το πιο προβληματικό όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, την οικονομική αυτονομία των γυναικών πρώτα απ' όλα. Η αλλαγή καθεστώτος έχει ως αποτέλεσμα ότι μετά από τις συζητήσεις μας μπορούμε να πούμε καθαρά ότι το σημερινό σύστημα των πανεπιστημίων δεν παράγει στελέχη που μπορούν να προσαρμοστούν στην αγορά. Ανάγκη λοιπόν προσαρμογή των ε, εκπαιδευτικών προγραμμάτων των πανεπιστημίων για τα σημερινά δεδομένα τη αγορά. Ένα πράγμα το οποίο δεν βρήκα στην έκθεση την ε, θέση τη γεωργία ω τομέα προτεραιότητα με είναι ένα τομέα με εξαιρετικέ δυνατότητε και δεν έχει την προτεραιότητα στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισία, για παράδειγμα. Μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό όσον αφορά τι μικροπιστώσει. Πράγματι, και εγώ συμμερίζομαι την άποψη τη κυρία Συγγήτρια ότι επί τόπου είδαμε γυναίκε που χρησιμοποίησαν τη ε, μικροπίστωση για να προχωρήσουν. Αυτό που μου δημιουργεί ερωτήματα είναι το επιτόκιο του 40%, δηλαδή παίρνουν μια πίστοση και πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια δεύτερη για να πλώσουν την πρώτη και μια τρίτη για να πλώσουν τη δεύτερη. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτά τα επιτόκια, τα υψηλά επιτόκια επιτρέπουν τελικά στις γυναίκες να είναι αυτόνομες αρκετά. Και τέταρτο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πιστεύω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους μηχανισμούς στην περίπτωση της Θηνησίας ή ε, ε, διπλή αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Task Force για την Αίγυπτο μετά από τις συνεδρίες της 13ης-14ης Νοεμβρίου όσον αφορά εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος ώστε να κάνουμε πιο έντονο του τόνου όσον αφορά θεμελιώδεις αρχέ τη δημοκρατία. Να συντονίσουμε τις προτεραιότητές μα, κυρίω όσον αφορά τι εμπορικές σχέσεις, βασιζόμενοι στην ανάγκη επαφή με την πραγματικότητα σε αυτέ τι χώρε Και τέλο, κάτι που εγώ πάντα θέλω να αναφέρω, την παρακολούθηση των εκθέσεων των εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικά έγγραφα που μας επιτρέπουν να μην εκπλησώμεθα όταν στις επόμενες εκλογές αντιλαμβανόμαστε ότι ό,τι είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια δεν ακολουθήθηκε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ευθύνη όλων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που μένει πάρα πολύ λίγος χρονο τώρα στο τέλο, Αλλά έχετε το λόγο έτσι πολύ σύντομα, εάν το επιθυμείτε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου να είμαι πολύ σύντομο παρόλο που έχω κρατήσει δύο σελίδε σημειώσει, δεν θα αναφερθώ σε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια για αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση και επίσης θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι ο ειδικό ανταποκριτής τη Λέβη Άστον έχει σε ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα τα δικαιώματα των γυναικών, Προφανώ, Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Όπως αναφέρθηκε, ε, υπήρξαν κύματα στη χρονική εξέλιξη της ε, κατάστασης και σε ορισμένες περιπτώσεις ανασυχητικές εξέλιξεις. Έχουμε δει προσπάθεια αποκλεισμού των γυναικών από τομείς της πολιτικής ζωής. Έχουμε ε, δει επίσης την διάπραξη εγκλημάτων με ατιμορρησία είτε από παρακρατικές ομάδες είτε από τις δυνάμεις ασφαλείας της κρατικές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και θετικές εξελίξεις όπως επίσης αναφέρθηκε. Όσον αφορά τους ε, παρατηρητές της, ε, την αποστολή παρατηρητών στις εκλογές, είναι κάτι που γίνεται. Έχει αποσταλεί οδηγία στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει να αποστέλουν ε, παρατηρητές στις εκλογικέ διαδικασίες και να συμπεριλαμβάνουν τα πορίσματά τους στις αναφορές που αποστέλουν στις Βρυξέλλες αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε συνεργασία με την Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, να, την, την πρόληψη και την δίωξη των υπέτειων για ε, βία κατά των γυναικών καθώς επίσης, έχουμε, όπως αναφέρθηκε, έχουμε αναθεωρήσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία και σε αυτό το πλαίσιο, καθώς επίσης και στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών συνεργασίας, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα, όπως αναφέρει και διεξοδικά κότερα πρόσωπος της Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι Συνολικά, η υιοθέτηση τον Ιούνιο από το Συμβούλιο του νέου στρατηγικού πλαισίου και του προγράμματος δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς επίσης και ο διορισμός του κ. Λαμπρινίδη στη θέση του ειδικού ε, εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε με μεγαλύτερη μαχητικότητα την ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έχουμε δημιουργήσει την ομάδα δράσης για την Αίγυπτο το Νοέμβριο και θα προσπαθήσουμε μέσω αυτής να εντείνουμε τις προσπάθειες για την ισότητα των δύο φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών. Σε περιφερειακό επίπεδο τώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της αραβικού Συνδέσμου έχουν ε, εντείνει τη συνεργασία τους. Διεξήχθη μια σύνοδο μια διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών του Αραβικού Συνδέσμου και στην οποία καταλήξαμε σε μια ε, διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με την οποία δεσμεύονται οι χώρες του Αραβικού Συνδέσμου στην πλήρη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητα των δύο φύλων. Επίσης έχουμε υιοθετήσει το πρόγραμμα εργασιών για τα επόμενα δύο χρόνια που συμπεριλαμβάνει στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ισότητα των δύο φύλων. Ευαρπιστούμε ότι θα υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα εργασιών συνεργαζόμενοι με τοπικές οργανώσεις. Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη, αλλά Έχουμε μόνο 20, 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας. Γιατί συνεχίζει ο εκπρόσωπο της EAS. Ένα στοιχείο για τη συνεργασία με το Young Women που αναφέρθηκε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους. Έχουμε συνάψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με την υπηρεσία αυτή, στο οποίο αναφέρεται και το πρόγραμμα που αναφέρθηκε και προηγουμένως, το Spring Forward και δεν θα πω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Σα ζητώ συγγνώμη γιατί σε λίγο θα λήξει το ωράριο των διερμηνέων. Και όλοι θέλουμε να πάμε για το μεσημεριανό γεύμα. Λοιπόν, θέλω να σας ε, ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Εάν πρόκειται να φύγετε τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη, χρονιά που πέρασε και δίνω το λόγο στην κυρία Κώστα να ολοκληρώσει πάρα πολύ σύντομα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ σα εύχομαι κύριε Πρόεδρε ότι καλύτερο σε εσά και σε όλου του συναδέλφου. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αρμαλεντόντα από τη Γραμματεία τη Κομισιόν, τη Επιτροπής επειδή έκανε πολύ σημαντικό έργο, πολύτιμο και το γεγονό ότι πήγαμε μαζί στην Τινησία Μα βοήθησε να έχουμε μια κοινή βάση. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλου του συναδέλφου, απλά κάποια σημεία εντάχει. Όσον αφορά ειδικότερα τη συνάδελφο κυρία Κράτσα, ένα πράγμα έχω υπογραμμίσει πολύ το θέμα της υποστήριξης και των γυναικών του Ισλάμ που εμπλέκονται σε αυτή τη δύσκολη επιδίωξη του καθορισμού της σχέσης μεταξύ Ισλάμ και Δημοκρατίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όπως είπε η συνάδελφος Ζαμπόσκα η κατάσταση αυτή αλλάζει κατά κύματα και μεταβάλλεται διαρκώς. Πρέπει Πρέπει να έχουμε διαρκώς υπόψη μας ε, τα επιτέγματα που συσσωρεύονται σιγά σιγά μέσα αυτών των διαδικασιών. Είναι πολύ σημαντικό το έργο της ε, συνέλευσης ε, για τη Μεσόγειο και ο ρόλος των βουλευτών σε αυτή τη συνέλευση και ήθελα να υπογραμμίσω και όλες αυτές τις νέες συμφωνίες που έχουν γίνει και με τον Αραβικό Σύνδεσμο και στο πλαίσιο διμερών σχέσεων με τις γυναίκες που έγιναν μετά από την παρουσίαση της εκθεσής μου. Ήθελα να πω ότι σύμφωνο στο να συνεχιστεί ε, αυτό το ζήτημα κατά του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Πιστεύω, ότι μάλλον συμφωνώ απόλυτα, όπως είπε η συνάδελφος κυρία Κράτσα και άλλοι συνάδελφοι, το ζήτημα ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στο διαθρησκευτικό διάλογο μεταξύ γυναικών στην Αίγυπτο υπάρχουν και οι κόπτες Υπάρχει μεγάλη, μεγάλος κίνδυνος μη σεβασμού της θρησκευτική ελευθερίας και των γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν εγώ υποστηρίζω το διαθρησκευτικό διάλογο μεταξύ των γυναικών και διάλογο μεταξύ των γυναικών και εντό των νέων ίδιων συνταγματικών διαδικασιών. Η Συρία δεν περιλαμβάνεται στην περίμετρο αυτή τη έκθεση. Τελευταίο πράγμα, η συνάδελφο Γκάμπριλ ειδικότερα και ο συνάδελφο Γκούσταυσον, συγγνώμη, δύο σημεία όπου μεταξύ πολιτικών και δημοκρατικών διαδικασιών πρέπει να κάνουμε διάκριση. Δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν τους πάντες. Και οι πολιτικές φυσικά. Θα βρούμε τον τρόπο στη συνάδελφο Γκάμπριελ. Η Γεωργία αναφέρεται. Σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί. Διότι είδαμε άμεσα στην νησία πόσο σημαντικό είναι και το ζήτημα των... της υπαίθρου όπου πρέπει να ακούσουμε το κόδωνα του κινδύνου όπως είπατε για να κλείσω, το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε μορφή συνεργασία και υποστήριξη τη χειραφέτηση των γυναικών. Δηλαδή, ανεξαρτησία να την ενισχύσουμε πολιτικά, κοινωνικά, σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα οικονομικά. Και για τις μικροπιστώσεις, ε, γι' αυτό ανέφερα ότι η Παγκοσμία Τράπεζα θα μπορούσε να ε, ορίσει ένα πρόγραμμα ταμείων εγγύησης που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα, όπως είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και λυπάμαι. Προθεσμία 15 Ιανουαρίου 17.00. 19 Φλεβάρι ψηφίζουμε και πριν να κλείσω να πω ευχαριστώ σε όλα τα μέλη, σε όλοι που συνεργαστήκανε πολύ καλά. Ευχαριστώ τους συμβούλους εδώ, τους συνεργάτες, τους πολιτικούς. Επίσης, να ευχαριστήσω τη συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και όλους τους οργανισμούς με τους οποίους είχαμε τη δυνατότητα και φυσικά να ευχαριστήσω τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ξεκουραστείτε, το χρειάζεται. Και τέλος, αλλά όχι ελάσσονος σημασίας, να, να εδώ ε, τη γραμματεία μου για όλο το έργο που έχουν καταβάλει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και καλά Χριστούγεννα. Και καλή χρονιά φυσικά. Γεια σας.